Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε με, την ε, Επιτροπή, τη δική μας. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των ε, συντονιστών. Σημείο 2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σε σχέση λοιπόν με την πρώτη εκδοχή της ημερήσιας διάταξης που σας εστάλει την περασμένη εβδομάδα υπάρχει μία διαφορά. Υπάρχει ένα αίτημα. Η έκθεση, η ψήφιση της έκθεσης ε, για τα αποθέματα βαθεών υδάτων να ε, μεταφερθεί, να αναβληθεί μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία για τις τροπολογίες. Και το σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης θα αντικατασταθεί, θα έρθει πιο νωρίς δηλαδή, θα ε, αλλάξει θέση. Η ανταλλαγή ε, απόψεων με πρόσωπο της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται όσον αφορά την Ισλανδία και τις Φερόες νήσους θα συζητηθεί σήμερα το πρωί και το 10 ε, αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις θα συζητηθεί το απόγευμα. Το 11 λοιπόν στη θέση του 10 και το 10 στη θέση του 11. Ο κύριος Αρσένης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόταση ήταν να γίνει στις 4 Νοεμβρίου. Η αναβολή να πάει για τις 4 Νοεμβρίου δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Δεν υπάρχει αντίρρηση από πλευρά μου. Δεν μου το είχαν πει ότι ήταν για τις 4 Νοεμβρίου. Αλλά ε, τώρα το έχετε μεταθέσει χρονικά για τις 4 Νοεμβρίου. Πολύ ωραία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν δεν θα ψηφίσουμε την έκθεσή σας σήμερα. Κύριε Λάβιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγκρίν, αφού είμαστε στη φάση έγκρισης της ημερησίας διάταξης, σας ε, ζητώ να επιτρέψετε στην νομική υπηρεσία να παρουσιάσει τη νομική γνωμοδότηση που λάβαμε χθες το βράδυ σε σχέση με την πολιτική, την αλλιευτική και τη συμφωνία επ' μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυριμπάτη, την οποία θα ψηφίσουμε άλλωστε ε, την έκθεση αυτή ε, τώρα αμέσω. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν πριν περάσουμε στην ψηφοφορία να ακούσουμε τη νομική υπηρεσία, να δεχθούμε ερωτήσεις και μετά να αποφασίσουμε πώς θα τοποθετηθούμε. Ο Πρόεδρος. Καλώς. Αυτό το οποίο προτείνεται λοιπόν είναι να συμπεριληφθεί ένα νέο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή συζήτηση για το θέμα αυτό. Διότι άλλη δυνατότητα είναι η εξή. την παρουσίαση της έκθεσης όλοι πήραν όλες τις πληροφορίες και μπορούσαν να τις διαβάσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να ξέρω και να καταλάβω τι προτείνεται. Πριν από την ψηφοφορία να κάνουμε ένα μικρό γύρο εξηγήσεων ή ερωτήσεων ή θέλετε να συμπεριλάβετε νέο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Η κυρία Ρόντους. Για την ψηφοφορία για τα ε, βαθαία είδη. Μπορώ να μιλήσω. Αν κατάλαβα καλά, προτείνετε κύριε Πρόεδρε, να γίνει ψηφοφορία όταν θα υπάρξει συμφωνία. Περίεργη η διαδικασία αυτή. Πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένη προθεσμία και να πούμε ότι εάν μέχρι τότε υπάρχει συμφωνία, καλώς. Γι' αυτό προτείνουμε να εμείνουμε στις 4 Νοεμβρίου. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε, δεν πρότεινα αυτό. Ως προς το κυριμπάτι να σας πω τι είπα. Ε, υπάρχει μια συμφωνία η οποία λέει ότι μετα... θα μετατίθεται η ψηφοφορία ε, την περασμένη συνεδρίαση που έπρεπε να την ψηφίσουμε, γιατί θα έπρεπε να ζητήσουμε ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Ε, και ότι αυτό θα το ψηφίσουμε σήμερα, είτε υπάρξει είτε όχι, συμφωνία νομική. Τώρα, η πρόταση ε, του μέλους ήταν να ε, γίνει συζήτηση σχετικά με την έκθεση. Και τη ρωτώ, θέλει να μπει καινούριο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή συζήτηση για την νομική έκθεση ή πριν από την ψηφοφορία να κάνουμε μόνο μια μικρή ανταλλαγή απόψεων. Η κυρία Λέβιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προτείνω να ακούσουμε μια σύντομη παρουσίαση από την νομική υπηρεσία και όσοι συνάδελφοι θέλουν να μπορέσουν να θέσουν και τις ερωτήσεις τους πριν την ψηφοφορία. Καλώ, η κυρία Φράγα παρακαλώ. Ναι, λοιπόν θα μιλήσω εξ ονόματος της ομάδας μου και θα πω ότι εμείς περιμένουμε την ψηφοφορία. Αυτό που είχαμε συμφωνήσει και ξέραμε ότι ήταν το συμφωνηθέν ήταν να ψηφιστεί όλο αυτό το πράγμα σήμερα. Έχουμε πάρει την έκθεση της νομικής υπηρεσίας, όλοι την έχουμε διαβάσει. Επομένως ο καθένας πράττει αναλόγως. Ε, και μάλιστα η νομική έκθεση δεν λέει τίποτα το οποίο να είναι αντίθετο με αυτή τη γραμμή πλεύσης. Νομίζω ότι τα μέλη που έχουν διαβάσει την έκθεση της νομικής υπηρεσίας μπορούν να ψηφίσουν εν πλήρη γνώση του περιεχομένου της έκθεσης της νομικής υπηρεσίας. Μπορούμε να κάνουμε μια μικρή συζήτηση και να υπάρξουν εξηγήσει για την έκθεση, αλλά από τη δική μου ομάδα δεν έχουμε καμία αμφιβολία και μπορούμε να περάσουμε μέσα στην ψηφοφορία. Ο κύριος Αντεπρεσέδο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τι είχαμε συμφωνήσει όλοι εμείς να ψηφίσουμε σήμερα και μάλιστα στην ομάδα εργασίας των σοσιαλιστών ε, πριν πάρουμε το περιεχόμενο της νομικής έκθεσης είχαμε συμφωνήσει να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο πριν περάσουμε στην ψηφοφορία να μας δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις και κάποιες εντυπώσεις για το περιεχόμενο της έκθεσης της νομικής υπηρεσίας. Ε, αυτό είναι αυτό που θέτω υπόψη σας γιατί αυτό είναι αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Η κυρία Ρόντις παρακαλώ. Και εγώ νομίζω ότι αυτό που είπε ο Αντολίν είναι σωστό. Θα μπορούσαμε σήμερα να το συζητήσουμε και σήμερα να ψηφίσουμε. Αυτό είναι σαφές. Μπορούμε να το κάνουμε. Προηγουμένως ε, ε, μίλησα για τα βαθαία είδη και εκεί θέλω να γίνει ψηφοφορία στις 4 Νοεμβρίου. Πρόεδρε, συγγνώμη, κύριε Ντέιβις, Πρόεδρε, μου λένε ότι το έγγραφο μοιράστηκε χθε. Από ποιον, με email ή διαζώσεις. Δεν το είδαμε πουθενά για να το διαβάσουμε. Λοιπόν, κύριε Ντέιβις, δεν θα αλλάζουμε κάθε φορά τα κριτήρια ψηφοφορίας. Εδώ ομόφωνα αποφασίσαμε ότι θα ζητήσουμε έκθεση από την νομική υπηρεσία. Συγγνώμη κύριε Ντέιβις, περιμένετε να ολοκληρώσω. Είχαμε λοιπόν συμφωνήσει ότι θα ζητήσουμε έκθεση από την νομική υπηρεσία και είτε βγει είτε δεν βγει, γιατί δεν ξέραμε αν θα υπήρχε, και θα, θα υπήρχε έκθεση από την νομική υπηρεσία εγκαίρως, ότι θα ψηφίζουμε σήμερα. Τελικά βγήκε η έκθεση χθε το απόγευμα πέντε και κάτι και στάλθηκε με email σε όλα ανεξα... ανεξαιρέτως τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με τον ίδιο τρόπο όλοι την πήραμε την έκθεση αυτή χθες και θέλω να τονίσω και το εξής. Τι έχουμε συμφωνήσει, ότι ανεξαρτήτως έκθεσης ή μη έκθεσης, αυτό το θέμα θα το θέσουμε προς ψηφοφορία σήμερα. Τώρα μπορείτε να μιλήσετε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μα είναι μόνο ένα το σημείο στην ημερήσια διάταξη, οι ψηφοφορίε. Μα είπαν να έρθουμε στι 9.30 γιατί θα ψηφίσουμε στι 10.30. Παρακαλώ, κάνετε τι ψηφοφορίε και μην επιτρέψετε άλλη συζήτηση. Ο κύριος, ε, κύριε Higgins, να σα πω ότι δεν σας καλέσαμε στις 9.30 για να ψηφίσετε. Ε, σας καλέσαμε στις 9.30 για να συζητήσουμε και να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και ακριβώς σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Λυπάμαι που βιάζεστε, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε, αλλά αλλά εγώ θέλω οι νομικοί μα σύμβουλοι να μα κάνουν μια δίλεπτη ανακεφαλαίωση για το κατά πόσον ή όχι πρέπει να ψηφίσουμε για αυτή τη συμφωνία ή όχι. Κατά τη δική του νομική άποψη, προπτική. Ευχαριστούμε, κύριο Στίβενσον. Ναι. Θέλω να συμφωνήσω με τον κύριο Χίγκιν όμω, πρόεδρε. Τα έχουμε διαβάσει κατά λεπτό. Δεν θέλετε να υπάρχει αντίφαση με την προηγούμενη εκδοχή που, μας, που είχαμε ήδη δει. Εάν η νομική υπηρεσία πάρει το λόγο, θα χρειαστεί ένα δεκάλεπτο και μετά όλοι θα θέλουν να θέσουν και ερωτήσει. Έχουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση κατά τα άλλα στι 10.30, οπότε πρέπει να ψηφίσουμε. Τα έχουμε ξανασυζητήσει όλα αυτά. Είχαμε ζητήσει νομική γνωμοδότηση. Τη διαβάσαμε, τα ξέρουμε, ε, τώρα πρέπει να ψηφίσουμε. Bien. Pues ya está... Καλώς. Λοιπόν, το θέμα έχει συζητηθεί. Εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη έτσι όπως είναι γιατί δεν τίθεται κανένα θέμα ε, διαφοροποίησης της. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ αφήστε με να τελειώσω και μπορεί να σας καλύψω. Εν πάση πτώση κυρία Ρόντους πείτε μου. Με συγχωρείτε. Θαύμασα Πώ εξηγήσατε στον κύριο Χίκη στον τρόπο εργασία μα. Νομίζω πω εξηγησατε στον κυριο χιγκιν τον τροπο εργασια μα νομιζω πω ηταν μια πολύ δημοκρατική προσέγγιση. Πολύ καλά. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να δράσουμε. Η κυρία Λεβίν ζήτησε να το συζητήσουμε. Εγώ το υποστήριξα. Ο Chris Davis επίσης το υποστήριξε. Δεν είναι δυνατόν να μην είναι δυνατόν στην Επιτροπή μας να πάρουμε 10 λεπτά για να συνηθίσουμε ένα θέμα όταν χρειαζόμαστε 10 λεπτά για να συζητήσουμε εάν θα το συζητήσουμε. Με συγχωρείτε αλλά δεν καταλαβαίνω. Δεν πρόκειται περί αυτού, κυρία Ρόντους. Θα το, αν με αφήνατε θα το είχα λύσει το θέμα είτε σας αρέσει τι λέει ο κύριος Χίγγινς είτε του κυρίου Χίγγινς του αρέσει τι λέτε εσείς ή όποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, μιλούμε για την ημερήσια διάταξη η οποία έχει υποστεί τις αλλαγές που έχουμε πει. Το μόνο είναι ότι αφαιρείται το σημείο για τα βαθαία ύδατα, δεν το ψηφίζουμε σήμερα την έκθεση του κυρίου Αρσένη και το 11 πάει στη θέση του 10 και το 10 πάει στη θέση του 11. Αυτές είναι οι μόνες αλλαγές. Τώρα μπορεί να γίνει μια συντομότατη ανταλλαγή από απόψεων πριν από την ψηφοφορία του Μπάτη και οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι το υποστηρίζουν αυτό, έχουν την πλειοψηφία έναντι των μελών του ΕΛΚ, επομένως συμφωνούμε. Μια συντομότατη, επαναλαμβάνω, ανταλλαγή απόψεων θα γίνει για τα του Κυριμπάτη. Υπάρχει έκθεση, δεν θα την εξηγήσει κανείς, ε, όποιος θέλει τη διαβάζει. Άλλο είναι μια συγκεκριμένη διευκρινιστική ερώτηση, και αυτό θα το επιτρέψω, και άλλο είναι η συζήτηση περί της ε, γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας. Όποιος δεν θέλησε δεν τη διάβασε και όποιος θέλει ας τη διαβάσει. Και τέλος, πάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Λοιπόν, το είπα και στην συνεδρίαση των συντονιστών. Θα λάβετε πρόσκληση για ένα σεμινάριο για την εφαρμογή ε, και την καλύτερη λειτουργία της ε, κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Μπορείτε να στείλετε βοηθό. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Το σημείο 5 λοιπόν αναβάλλεται και γι' αυτό περνούμε στο σημείο 6. Το ανώτατο ένα λεπτό θα δώσω στον, σε κάποιον από εσά, εάν θέλει να πάρει το λόγο για κάποια διευκρινιστική μόνο ερώτηση και τίποτα άλλο. Κύριε Ντέιβις, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βρήκα το μέλη του κ. Χόπκινς, είδα του τρει τελευταίε παραγράφους, το τέλο του και δεν τις καταλαβαίνω. Ο κ. Χίγκιν μπορεί να μου τι εξηγήσει. Αν θέλει τόσο πολύ να ψηφίσουμε άμεσα, να μου πει τι καταλαβαίνει από την νομική ερμηνεία τη υπηρεσία. Διότι αν εδώ δεν είμαστε σώμα εκλεγμένων αντιπροσώπων, τι είμαστε, τι δημοκρατία υπάρχει. Είμαστε ανεπαρκεί νομοθέτε. Ε, ο νομοθέτη θέλει να ξέρει τι ακριβώ σημαίνει η νομική πράξη που ψηφίζει. Με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω αυτά τα δικηγορίστικα λόγια, Πρόεδρε. Κάποιο που ξέρει από νομική να μου εξηγήσει και από δίκαιο. Ποιε είναι οι επιπτώσει δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ μια τέτοια συμφωνία. Θα ψήφιζα μάλλον υπέρ τη συμφωνία, αλλά τώρα θα καταψηφίσω γιατί δεν καταλαβαίνω ποιε θα είναι οι επιπτώσει, ποιε θα μπορούσαν να είναι. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντέβι, τώρα τι καταλαβαίνει ο καθένα ε, από αυτά που διαβάζει, γι' αυτό έχουμε του βοηθού και του συμβούλου μα. Και ο καθένα είναι ελεύθερο να καταλάβει ό,τι νομίζει. Αλλά η κυρία Ρόντου τι θέλει το λόγο. Συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν θα ήθελα να ερμηνεύσω, θα ήθελα να μου πει η νομική υπηρεσία εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι νομικοί λόγοι για να υποστηρίξουμε αυτή τη συμφωνία ή αν είναι κάτι το ασαφές και θα εξαρτηθούν όλα από τον τρόπο εφαρμογής. Θα ήθελα να μάθω τι θα την κάνουμε αυτή τη συμφωνία. Αλλιώς δεν μπορώ να αποφασίσω σήμερα. Ευχαριστώ να πω στον κύριο Χιγκίνς ότι λυπάμαι που έχει προκύψει έτσι η κατάσταση. Εγώ ήθελα η γραμματεία να το συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη, να προβλεφθεί ως σημείο, το ζήτησα. Αλλά τέλος πάντων, η ερώτησή μου προς την νομική υπηρεσία είναι το, η εξή. Για τη συμπερίληψη για τη συντήρηση και για τα μέτρα συντήρησης και διαχείρισης το 2012 και τη συμπεριλήψη των μέτρων αυτών που δεν υπάρχουν στο πρωτόκολλο, πώς θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο ισχύον πρωτόκολλο. Διότι όπως ε, παρουσιάζεται αντιφάσκη με τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συμβαλόμενου μέρους στο WETFC. Η... Θα πρέπει να μας ε, εξηγήσει η νομική υπηρεσία, όχι βέβαια την έκθεση που όλοι τη διαβάσαμε, αλλά να μας πει, ε, να μας δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα, να απαντήσω στις δύο ερωτήσεις της κυρίας Ρόντουστ και της κυρίας Λέβιν. Η κυρία Ρόντουστ ρώτησε ακριβώς εάν υπάρχει κόλλημα για την σύναψη του πρωτοκόλλου από νομικής ε, σκοπιάς ή αν θα μπορούσε να ερμηνευτεί διαφορετικά το πρωτόκολλο προς την νομιμότητά του ή όχι. Η απάντηση είναι προς τη δεύτερη ε, επιλογή. Δηλαδή συμπεραίνουμε ότι το πρωτόκολλο αυτό καθε αυτό μπορεί να είναι νομικός αποδεκτό με την παράγραφο 37 του κειμένου μας αρκεί να ερμηνεύεται βάσει και σύμφωνα με το ισχύοντα μέτρα συντήρησης και διαχείρισης. Εν προκειμένου με τους αριθμούς του 2012, διότι στο κείμενο του πρωτοκόλλου υπάρχει μια σαφής μνήα, όπως ε, υποδεικνύουμε στην παράγραφο 19, ότι οι αλλιευτικές ευκαιρίες πρέπει να οριστούν βάσει των όριων που έχει καθορίσει η Επιτροπή Δυτικού και Ανατολικού Ατλαντικού ε, μέτρα συντηρήσεω και διαχείριση και όχι υποχρεωτικά βάσει του 2008 αριθμό 1. Αυτό έχει καταστεί παροχημένο, ξεπερασμένο, διότι έχει ουσιαστικά καλυφθεί από το επόμενο πρωτοκόλλο. Και για το ερώτημα της κυρίας Λέβιν, πώς αυτή η δεύτερη εκδοχή των μέτρων συντήρηση και διαχείριση του 2012 μπορούν να συμπεριληφθούν στο ισχυρό πρωτόκολλο, η απάντηση εδώ είναι με ερμηνευτικές μεθόδους. Δηλαδή και πάλι ε, συμπεραίνουμε στις παραγράφους 32 και 35 ότι βάσει των εδαφείων B και C, Β και Γ, το πρωτόκολλο μπορεί να συναυθεί υπό τον όρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει προσπάθειες να εξασφαλίσει ότι στην πράξη αρχές του Κυριμπάτη εφαρμόζουν ε, τη συμφωνία βάσει των μέτρων διαχείρισης και συντηρήσεως που έχουν συμφωνηθεί. Δηλαδή ότι το δίκαιο γίνεται σεβαστό και από τις δύο συμβαλόμενες πλευρές. Βεβαίως, το θέμα της, ε, ε, πρα, της πρακτικής εφαρμογής του πρωτοκόλλου, δηλαδή αν αυτές οι συνθήκες θα εκπληρώνονται ή όχι, αυτό είναι κάτι που επίπτει στις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και Κυρίε και κύριοι βουλευτές. Ωραία. Θα σα δώσω το λόγο για ένα λεπτό, όχι για να αρχίσουμε συζήτηση, αλλά για να καταλάβουμε τι μα είπε η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλου, πολύ γρήγορα και πολύ συγκεκριμένα. Κατά την άποψή μα δεν αντιφάσκει καθόλου αυτό που ακούστηκε με αυτά που είπε σε προηγούμενε συζητήσει εδώ για το η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αν διαβάσετε τα συμπεράσματα τη εκθέση αυτή, είναι σαφέ ότι οι ελευθερικέ δυνατότητε ελευθερικέ μάλλον ευκαιρίε, ε, αναφέρονται στη σελίδα 8 του σημείου 38. Θα πρέπει να προβλέπονται για τη αλληλευτικά τη Ευρωπαϊκή και βάσει των ορίων που έχει ορίσει η Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ακριβώ μα λένε και οι αρχέ του κ. Μπάτη. Αυτό μα έχουν πει επανειλημμένω κατά τι διαπραγματεύσει και κατά τι μεικτέ επιτροπέ. Ε, το γεγονό ότι στο πρωτόκολλο υπάρχει ε, μια τέτοια μνήμα δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει το πρωτόκολλο. Ε, εφαρμόζεται με τη, με μετάφραση των διατάξεων αυτών καθημερινά σε μέρες. Έτσι ε, φαίνονται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους. Εφόσον α, είναι και αυτοί μέλη του DNA. Ε, οπότε αυτό ήθελα να καταστεί σαφές. Από νομική πλευρά βρίσκω ότι υπάρχει ένα σφαλματάκι. Διότι τα μέτρα συντήρηση που αναφέρονται εδώ είναι τα μέτρα που επιβλήθηκαν και πριν και μετά πριν αρχίσουμε να συζητούμε και να υπογράψουμε το πρωτόκολλο. Όμως το 2011 τα μέτρα αυτά, αυτά τα μέτρα του 2011 δεν αναφέρονται. Αυτό θέλω να έχω υπόψη τους όλοι. Ευχαριστώ. Δεν θα πάρει κανείς άλλο το λόγο. Θα ψηφίσουμε. Το πρωτόκολλο Ευρωπαϊκή Ένωση Κυριμπάτη για τις δυνατότητες αλληλείας. Έχετε όλη την κάρτα σας. Ωραία, να αρχίσουμε την παράγραφο 1. Τροπολογίες 1 και 2. Ενάρξη λήξη. Κάτι έγινε. Λοιπόν, άρχεται εκ νέου ψηφοφορία. Άρχεται. Λήξη. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. <clears throat> Τροπολογία 3. έναρξη. Οι σοσιαλιστές ψηφίζουν με μία ψήφο παραπάνω. Ωραία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται. Λήξη. εγκρίνεται. Τροπολογία 5 και 6 που είναι ταυτόσιμες. Άρχεται. Πέντε και έξι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Λοιπόν, ναι, ας ξαναρχίσουμε την ψηφοφορία, ξανακάνουμε την ψηφοφορία. Τροπολογίες 5 και 6. Άρχεται, πέρας, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τροποποιημένο σχέδιο, ε, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται, πέρας, Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται. Επόμενο θέμα. Κύριε Ντέβις, ε, ε, μας δίνετε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 3 κατά, 0 αποχές. Με συγχωρείτε. 18, 3, 0. Επόμενο θέμα. Είναι η γνωμοδότηση της κυρίας Τόμα συμβαστική 1 άρχεται πέρας εγκρίνεται τροπολογία 69 άρχεται πέρας Λοιπόν, πρέπει να ξαναρχίσουμε. Αν θέλετε να γίνει διανατάσεως, ε, γιατί άρχεται πέρας, για να δούμε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Άρχεται. Πέρας. Σας παρακαλώ ησυχία. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Ε, άρχεται. Πρόεδρε, πρέπει να δούμε τι έγινε με την ψηφοφορία μα Δεν βλύναμε τις ψήφου μας. Θα σα πω το αποτέλεσμα. 71 άρχεται. 71. Πέρας. 16-5. Εγκρίνεται. 72. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 18-3. 73 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 16-5. Να, θα γίνεται διανατάσεως διότι δεν ξέρω τι γίνεται. Τροπολογία 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.

18 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 α, εγκρίθηκε 77 υπέρ 77 κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ Δύο τμήματα, μάλιστα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τη συμβαστική τρία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 που είναι ίδια με 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά ε, κατά παρακαλώ εγκρίνεται 35 υπέρ Παρακαλώ ε, να σηκώνετε τα χέρια σας. Κατά αποχές εγκρίνεται. «163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ε, συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε τώρα την τροποποιηθής γνωμοδότηση. Λοιπόν, ε, πρέπει να έχουμε τον αριθμό των ψήφων ηλεκτρονικός. Λοιπόν, άρχεται. Τώρα πρέπει να έχουμε το ακριβές, τον ακριβή αριθμό. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Λοιπόν, άλλη μια φορά παρακαλώ. Πέρας. Δεκανέα υπέρ, δύο κατά, μηδέν αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τωμά. Εγκρίνεται. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης τροποποίηση του Πρωτοκόλου του 1224 διότι έχουμε ε, ε τροποποίηση του κανόνα στην κοινή ελευτική πολιτική. Η Επιτροπή ε, παρουσίασε την άποψή της το Μάρτιο, το συζητήσαμε τον Ιούλιο και η κυρία Τομάς θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης και τη δίνω το λόγο ευθύ αμέσως παρακαλώ. Και σας παρακαλώ επίσης να κάνετε ησυχία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα είμαι και αρκετά σύντομη. Θέλω να σας υπενθυμίσω το μοναδικό στόχο αυτής της έκθεσης είναι να υπάρξει συμμόρφωση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και αυτό ισχύει και για διάφορες άλλες εκθέσεις, τις οποίες έχουμε ήδη ψηφίσει. Είναι πιο εύστοχο αυτό και για να συμβαδίζει με τη νέα κοινή ελεκτική πολιτική. Θα έχουμε ένα νέο κανονισμό ελέγχου λοιπόν, οπότε δεν είναι τόσο σκόπιμο να προσπαθούμε να περάσουν ε, τροποποιήσεις ε, επί της ουσίας αυτή την έκθεση. Μιλάμε απλώς για μια λισαβονοποίηση. Απλώς να επιμείνω στον ε, ουσιώδη χαρακτήρα των exposed ελέγχων που προβλέπονται από τις κατεξουσοδότηση πράξεις, διότι όσο και αν έχουμε επανειλημμένω ότι αυτές οι πράξεις στην πραγματικότητα είναι πράξεις που εξοδοτεί το Κοινοβούλιο να κορυφούν ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, δεδομένης της φύσης των πράξεων αυτών που τις καθιστά ε, σημαντικές, εάν δεν υπάρχει εξπόστα έλεγχος του Κοινοβουλίου, θα βρεθούμε όχι να έχουμε εκχωρήσει κάτι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να ουσιαστικά να τις έχουμε παραχωρήσει ένα μέρος της εξουσίας μας. Ε, ως προς την ίδια την έκθεση, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι εκτελεστικές και οι κατεξοδοσόντες συμπράξεις κάνει τη σωστή διάκριση βάσει της συναπόφασης, αλλά πρέπει να δούμε ακριβώς τον ex έλεγχο ο οποίος επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να διευκρινίσει τι ακριβώ περιμένει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με συγχωρείτε, έχει πολύ θόρυβο δίπλα μου και είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί κανεί αυτό που μιλάει. Ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι μπορεί το Κοινοβούλιο να δώσει συγκεκριμένες συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τον τρόπο που θεωρεί ότι αυτές οι κατεξοδότηση πράξεις μπορούν να εφαρμοστούν. Ένα παράδειγμα, διότι είναι μέρος των ε, προσθήκων που πρότεινα στην έκθεση αυτή, ε, κατά πράξη που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαιρέσει τα σκάφη από την προθεσμία κοινοποίηση ε, πρόσθεσης που είναι 24 ώρες. Αυτή η εξαίρεση σήμερα στον κανονισμό ελέγχων όπως ε, ισχύει γίνεται ανάλογα με τον τύπο του σκάφους. Σκέφτηκα όμως ότι ο όγκος, για αυτό το είδος την εξαίρεση, η χωρητικότητα δηλαδή, ίσως να είναι ένα ε, ευστοχότερο κριτήριο. Δηλαδή, αν έχει κανείς να εκφορτώσει 100 κιλά ψάρια, θα έπρεπε να έχει περίοδο εκφόρτωσης ε, πιο μεγάλη, πιο σύντομη μάλλον από ότι αν είχε ελάχιστος τόνους να εκφορτώσει. Εδώ λοιπόν Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια-δυο τέτοιε προσθήκε ώστε να, υπάρχει, να υπάρχουν κάποιε περισσότερε ενδείξει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για να ολοκληρώσω. Δύο ακόμα στοιχεία, να Ε, πρότεινα αυτή η εξουσιοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ισχύει για μια τριετία. Αλλά δεδομένων όσων έλεγα για τον απαραίτητο εξπρόστα έλεγχο του Κοινοβουλίου, ως προς τις κατεξοδότηση πράξεις. Για αυτό το σκοπό πρότεινα εννέα μήνες πριν την εκπνοή της περίοδου να ετοιμάζεται έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αξιολογείται η χρησιμότητα των πράξεων υπό την έννοια της κοινή ελευτικής πολιτικής και του κανονισμού περί Τέλος και καταληκτικά, κατά την ανάγνωση αυτού του κανονισμού, προέκυψαν κάποιες απορίες. Αντιλήφθηκα ότι προβλεπόταν κάτι σαν κύρωση. Μια κύρωση που αντιφάσκει με τη Χάρτα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Μία από τις κυρώσεις δηλαδή που προβλέπει ο κανονισμός. Ουσιαστικά τιμωρεί σε περίπτωση παράβασης όχι τον ε, υπεύθυνο είτε τον καπετάνιο είτε τον πλειοκτήτη αλλά τιμωρεί το σκάφος. Αυτό σημαίνει ότι η τιμωριακή ρωσή δεν έρχεται να πλήξει αυτόν που είναι υπεύθυνο που την προκάλεσε, αλλά το σκάφος ε, σε περίπτωση κατάσκησης. Στη νέα όμως συνθήκη, τη συνθήκη ε, βάσει της οποίας εφαρμόζουμε τη λισαβονοποίηση. Εκεί ε, υπάρχει ως παράρτημα η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν μια παράπατη νομική αναφορά και ένα σημείο αναφοράς. Δεν βλέπω λοιπόν πώς αν θέλουμε να περάσουμε στην διάσταση της Λισαβόνας ε, και να ευθυγραμμιστούμε με αυτήν, πώς μπορούμε να έχουμε ένα κανονισμό που να αντιφάσκει με τη χάρτα, η οποία αυτή η ίδια έχει νομική ισχύ μέσω της συνθήκης. Γι' αυτό Ζήτησα από τον Πρόεδρο και φαντάζομαι ότι το είπατε αυτό στην ε, συνεδρία των συντονιστών να έχουμε μια νομική ε, διευκρίνηση εδώ. Δεν γνωρίζω εάν αυτό πώς να το πω διακόπτει και κάνει να παραλύσει η διαδικασία. Πιστεύω ότι η έκθεση μπορεί να ψηφιστεί και η διόρθωση να γίνει εκ των υστέρων. Όμως ε, Ήθελα να μου πείτε τι έγινε με αυτήν την νομική απορία και την διευκρινιστική απάντηση που ζητήθηκε. Μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μου έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Α, δεν σας είχα Συγγνώμη, κυρία Φράγκα, παρακαλώ. Λοιπόν, Ευχαριστώ καταρχάς την κυρία εισηγήτρια, την κυρία Τομάς για την έκθεση αυτή. Είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει πολύ λιγότερο από ότι ε, η συζήτηση για το κυριμπάτι. Υπάρχει ευθυγράμμιση και ενδεχομένως μπορεί να είναι και αρκετά ανιαρό. Και θα ακολουθήσω λοιπόν και εγώ σε αυτή την ανιαρή, ανιαρή γραμμή και να κάνω ορισμένα σχόλια για τις τροπολογίες. Πρώτον, Καταρχάς, στην ε, τροπολογία υπαριθμών τερία Νομίζω ότι είναι αμφισβητήσιμη η τροπολογία σας. Ο κανονισμός, έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή, αναφέρεται στα μικρά αλλιευτικά σκάφη στο άρθρο 5 ε, ως προς τις εγκρίσεις για την αλλιευτική δραστηριότητα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο μέλλον θα συνεχίσουν έτσι τα πράγματα. Ε, μπορεί να εξαφανιστεί αυτή η δράση ή να υποβληθεί σε περισσότερους όρους και προϋποθέσεις. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου μιλούμε για την ε, θέσπιση κανόνων να έχουμε ε, εκτελεστική πράξη και όχι κατεξουσιοδότηση πράξη. Αυτό είναι πολύ καλύτερο κατά τη γνώμη μου. Τώρα, στην τροπολογία υπαριθμού 4, γιατί μιλάει για τα πρότυπα που εμφανίζονται στο σημείο C. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό αυτό και συμφωνεί περισσότερο με τη διαδικασία της, τροπολογ... της επιτροπολογίας. Ως προς την τροπολογία υπαριθμών 6, συμφωνώ επί της ουσίας με το περιεχόμενό της, ωστόσο κάτι που έχω επαναλάβει στο Κοινοβούλιο είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την ευθυγράμμιση, θα πρέπει να μην παρεκκλίνουμε από την ευθυγράμμιση των κειμένων με τη συνθήκη και να μην μπαίνουμε σε θέματα επί της ουσίας. Και όμως, εσείς εδώ ακριβώς αυτό κάνετε. Ενώ θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε όλα τα κείμενα με τη συνθήκη, ε, μπαίνετε επί της ουσίας. Με αυτή την παρέκκληση θέτετε εσείς ένα θέμα επί της ουσίας και εγώ δεν συμφωνώ, το έχω πει επανειλημμένως, ότι δεν θα δεχτώ να μπαίνουν από το παράθυρο ε, για συζήτηση ζητήματα επί της ουσίας, όταν ο σκοπός μας είναι μόνο να ευθαγραμμίσουμε τα κείμενα. Τώρα, στη συνέχεια χρησιμοποιείται ένα νέο όρο, ε, όρο του όγκου. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ε, σε τι οφείλεται, μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Και στην τροπολογία υπαριθμών 8 δέχομαι να διατηρηθεί η πρωτοβουλία του κράτους μέλους, αυτό προτείνετε εσείς, όπως και υπάρχει στον υφιστάμενο κανονισμό, όμως καλύτερα να έχουμε εκτελεστική πράξη και όχι κατεξουσιοδότηση πράξη. Ε, ε, νομίζω ότι θα είναι πιο λειτουργικό το σύστημα έτσι. Στη συνέχεια ε, δεν συμφωνώ μαζί σας να μην εξαφανιστεί η Τεχνική και Οικονομική Συμβουλευτική Επιτροπή Αλίας. Το έκανε η Επιτροπή για να συνάδει το κείμενο με το νέο κανονισμό που θα χρησιμεύσει ως νομική βάση. Αλλά αφού δεν έχει αρχίσει να ισχύει αυτός ο κανονισμός, συμφωνώ να διατηρηθεί αναφορά σε αυτή τη Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή. Στη συνέχεια, στην τροπολογία 10, μιλούμε για την ανιχνευσιμότητα ή την ιχνηλασιμότητα. Εδώ τίθεται ένα πρόβλημα. Λέτε εσείς ότι το διαγράψατε αυτό το καταργήσατε γιατί έχει να κάνει με την κοινή οργάνωση αγοράς η οποία όμως δεν έχει αρχίσει να ισχύει ακόμα και εάν πρέπει συνεχώς να λέμε ότι θα κάνουμε ότι ό,τι και να κάνουμε πρέπει να συνάδει με το OCM, τότε θα πρέπει να αφαιρέσουμε πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει συνοχή ή θα αφήσουμε το κείμενο ως έχει ή αν θέλουμε να συνάδουμε με την ΩΣΕΜ θα διαγράψουμε και θα, θα αφαιρέσουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό μόνο. Τώρα, τροπολογία 13 και 14. Ε, μιλούν για θέματα επί της ουσίας. Δεν μπορώ να τις δεχτώ. Επί της αρχής είναι το θέμα. Τροπολογία 15 δέχεστε εδώ εσείς ε, την πρόταση της Επιτροπής ε, κατά τη διαδικασία της Επιτροπολογίας και υπάρχει αυτή η παρέκκληση για την τριετή περίοδο για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και εξουσιοδοτήσεις και ούτω καθεξής. Αλλά εγώ τους άλλους δεν συμφωνώ, δεν θεωρώ ότι όλες οι πράξεις θα είναι και πρέπει να είναι ε, κατεξουσιοδότηση. Επομένως μου δημιουργεί πρόβλημα η τροπολογία σας. Τώρα η 16. Δεν διαφωνώ αλλά νομικώς δεν ξέρω αν είναι εφικτό να ζητηθεί αυτή η λογοδοσία από πλευράς Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο πάντοτε ασκεί τον έλεγχο. Δεν είμαι κατά, αλλά ε, νομικά νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα εκεί και θα πρέπει να διευκρινιστεί. Τώρα, ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σας θέσω ένα ερώτημα που έχω ξαναθέσει αλλά δεν μου έχει απαντηθεί. Το 404 στερείται νοήματος με αυτόν τον κανονισμό. Θέλω να μου πείτε, το να αφαιρέσουμε ολόκληρα τμήματα από του ε, περιεχομένου, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτής της αφαίρεσης στο άρθρο 404. Ξέρω ότι όλα αυτά είναι πολύ ανιαρά. Δεν θέλω να κουράσω άλλο τους συναδέλφους. Έχει δουλέψει πολύ η κυρία Τομάς ως προς αυτό και γι' αυτό δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα. Ήδη αυτά που υπόθηκαν έχουν ε, ε, προλάβει πολλά από αυτά που ήθελα και εγώ να πω και εγώ πιστεύω ότι μια διαδικασία λισαβονοποίησης πρέπει να περιορίζεται σε αυτό. Συμφωνώ για διάφορα θέματα που ανέφερα, ιδιαίτερα την τροπολογία 3 που είναι θέμα ουσίας, αλλά και την τροπολογία 6 για μένα αυτό που είναι σημαντικό είναι η 6 και η 13. Η 13 γιατί γιατί η αλλαγή του συστήματος ε, πόντων είναι ένα πολύ βασικό θέμα. Καταλαβαίνω ότι οι μηχανισμοί θα μπορούσαν να δώσουν συνέπεια στο σύστημα και μέσω της λισαβονοποίησης να το αλλάξουμε αυτό ανοίγει ένα παράθυρο που νομίζω ότι είναι δύσκολο. Αυτό που μας ε, ανησυχεί είναι η δυνατότητα που δίδεται να αρχίσει μια συζήτηση που δεν είναι αυτή τη στιγμή σκόπιμο να την ε, ανοίξουμε. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να περιοριστούμε στη λισαβονοποίηση και το θέμα ουσίας θα το συζητήσουμε αλλού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα. Δεν μου ζήτησε άλλο το λόγο. Η Κομισιόν, ο κύριος Πένας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστούμε την κυρία Τομά για την έκθεση, της τροπολογίας να σας ενημερώσω ότι γενικά η Κομισιόν συμφωνεί με την κατανομή των πράξεων ε, που προτείνει η κυρία Τομά διότι η ερμηνεία της συμπίπτει ε, σε μεγάλο βαθμό με το ποια θέματα πρέπει να είναι κάτω εξουσιοδότηση και ποιες διατάξεις πρέπει να ε, μετατραπούν σε εκτελεστικές πράξεις να αναφέρω ορισμένα θέματα που ανέφερε και η κυρία Τομάς και η, κυρία Φράγκα και η κυρία Φράγκα και ο κύριος Ζωμέβα. Είναι σαφές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι αποκλειστικός στόχος είναι ο κανονισμός ελέγχου να προσαρμοστεί στη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν είναι σκόπιμο σε αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε συζήτηση για θέματα ουσίας. Ιδιαίτερα εάν τα θέματα αυτά γιατί αυτό μπορεί να προκύψει από κάποιες τροπολογίες, μπορεί να ε, αποδυναμώσουν τον ε, κανονισμό ελέγχου. Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι το Κοινοβούλιο θέλει να ελέγχει αυτές τις πράξεις, παρόλα αυτά, από την επόμενη χρονιά, όταν θα εγκριθεί ο νέος βασικός κανονισμός της κοινή ελευτικής πολιτικής με βάση το 46, το άρθρο 46, θα δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασία για την εφαρμογή των κανονισμών ελέγχου και αυτή η ομάδα εργασία θα συμπεριλάβει και το Κοινοβούλιο όπως ακριβώς πρότεινε το Κοινοβούλιο στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου είναι αυτή η ομάδα εργασία. θα αρχίσει να λειτουργεί από την επόμενη χρονιά με στόχο προφανώς να καλέσει και το Κοινοβούλιο ούτω ώστε να διαδραματίσει το ρόλο που το αναλογεί για τον έλεγχο της πολιτικής ελέγχου. Επί της ουσίας συμφωνούμε δηλαδή ότι το Κοινοβούλιο θα παίξει σημαντικό ρόλο εφόσον στα πλαίσια του, κανονισμού, του βασικού κανονισμού θα αρχίσει να λειτουργεί αυτή η ομάδα εργασία. Θα έχει λοιπόν βήμα για να εκφράσει τις απόψει του. Επίσης, το εάν και κατά πόσο θα υπάρξει έκθεση για την εφαρμογή των κατεξουσιοδότησης πράξεων μας φαίνεται πρόωρο να αρχίσουμε ήδη να ε, συζητάμε ενδεχόμενο τέτοια έκθεση για δύο λόγου. Όπω ξέρετε, ο κανονισμό ελέγχου, ελέγχου δεν έχει εφαρμοστεί πολύ καιρό και μία από τι διατάξει του και ορισμένε διατάξει του ακόμη δεν έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Τώρα αρχίζουν να εφαρμόζονται, διότι σταδιακά εφαρμόζεται. Άρα μέχρι στιγμή ούτε καν όλε οι διατάξει δεν ισχύουν. Και όπω ξέρετε, ο κανονισμό προβλέπει μία γενική αναθεώρησή του και τη εφαρμογή του το 2015. Οπότε να προσθέσουμε και άλλες υποχρεώσεις χορήγησης πληροφόρησης για την εφαρμογή πριν από αυτή τη γενική έκθεση που θα έχουμε το 2015 νομίζουμε ότι είναι περιπλοκή που επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θεωρώ ότι αιτιολογείται. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι πρέπει να αναλύσουμε το σύνολο ε, της εφαρμογής του κανονισμού, όχι μόνο τον κατ εξοδότης συμπράξεων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την κυρία Τωμά που λέει ότι πρέπει η Κομισιό να αποτιμήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Συμφωνούμε. Αλλά νομίζουμε, κυρία Τωμά, ότι πρέπει να το δούμε σφαιρικά στα πλαίσια της εφαρμογής του κανονισμού, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του που προβλέπεται για το 2015 και όπου το Κοινοβούλιο θα παίξει σημαντικό ρόλο. Σύντομα τώρα, να αναφερθώ στην τροπολογία 13 για το σύστημα πόντων. Είναι ένα νέο στοιχείο του κανονισμού ελέγχου. Επιτρέψτε μου να πω ότι πολύ πρόσφατα άρχισε να ισχύει όλα τα, μέτρα, τα κράτη-μέλη δεν έχουν μπορέσει ακόμη να το εφαρμόσουν. Είναι νέο στοιχείο. Είναι σε φάση εφαρμογής. Τώρα να το τροποποιήσουμε ενώ ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί πλήρω ε, ε, είναι πρόωρο κατά τη γνώμη μας διότι στην πρόταση που μας κάνει η κυρία Τομά θεωρούμε ότι υπάρχουν στοιχεία που θα αποδυνάμωναν τον έλεγχο το σύστημα λοιπόν αυτό των πόντων δεν πρέπει να αφορά και να εφαρμόζεται μόνο στον ε, πλειοκτήτη αλλά και στον εφοπλιστή που είναι κάτοχος της άδειας αλίευσης. Συμφωνούμε με την κυρία Τομά ότι αυτή η νομοθεσία, όπως κάθε νομοθεσία, πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με την χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Βεβαίως, φυσικά, συμφωνούμε. Αλλά αυτή η διάταξη να εφαρμοστούν οι πόντοι και στον κάτοχο της άδειας, κατά τη γνώμη μας, δεν αντιβαίνει θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί πρέπει να σας εξηγήσω κάτι σημαντικό. Το σύστημα πόντων προσπαθεί να αποθαρρύνει την κακή συμπεριφορά. Αλλά όχι μόνο του καπετάνιου. Ξέρουμε από πολιετή πείρα ότι αυτή η κακή συμπεριφορά του καπετάνιου έχει επιβληθεί από τον εφοπλιστή, από τον κάτοχο της άδεια. Γι' αυτό το σύστημα πόντων πρέπει να εφαρμόζεται για να αποθαρρύνει τις ε, καταχρήσεις και στον ε, κάτοχο της άδεια αλίευσης. Είναι θέμα λοιπόν ε, γενικής προσέγγισης. Γι' αυτό εμένουμε ιδιαίτερα. Δύο θέματα που έθεσε η κυρία Φράγα η ιδέα του φέθε. Το να μην προβλέπετε κάτι τέτοιο οφείλεται στο ότι η Κομισιόν με βάση το βασικό κανονισμό δεν θέλει το SFTS να είναι η μόνη πηγή ε, επιστημονικής πληροφόρησης. Ε, η κοινή ελευτική πολιτική υποβάλλει πολλές ερωτήσεις στους επιστήμονες Δεν θέλουμε λοιπόν ε, ε, και άλλες ε, εκθέσεις. Πρέπει να βασιστούμε στην επιστημονική πληροφόρηση που μας δίνει αυτός ο φορέας, αλλά και άλλοι φορείς. Δεν είναι σκόπιμο λοιπόν να υπάρχει επικάλυψη της εργασίας του SSTF που είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο, με την εργασία που θα μας δίνουν άλλοι ε, φορείς για τον κανονισμό για τις αγορές τώρα. Λοιπόν, συμφωνούμε ότι στο πλαίσιο της έγκρισης του κανονισμού της κοινή οργάνωσης αγορών θα υπάρξει μια δήλωση των δύο κλάδων της νομοθετικής εξουσίας να κάνουν αίτηση στην Επιτροπή να εξετάσει το θέμα αυτό και βέβαια για αυτό το θέμα η Επιτροπή θέλει, θα χρειαστεί μία κατεξοδότηση πράξης. Αυτό βέβαια θα είναι απέτηση των συνομοθετών στα πλαίσια της απόφασης για τον κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την εξοδότηση γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε αυτό που θα μας ζητούν στη δήλωση οι συνομοθέτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πένας. Νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τομάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ελπίζω ότι τα σημείωσα όλα σωστά. Μπορεί να υπήρξαν κάποιες αυλεψίες, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε και διμερώς και στην, ε, στις συνεδριάσεις των σχεδόν συγκητών. Κατά πρώτον, για τις τροπολογίες 3 και 4. Πρόκειται για μία μετατροπή βάσει των όσων ε, λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η αρχική έκφραση ήταν αμφίσιμη και επέτρεπε παρερμηνίες. Δεν θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν τέτοιες παράλληλες ερμηνείες. Δεν υπάρχει αλλαγή στην ουσία. Τροπολογίες 7 και 6. Εδώ η ίδια η φύση των κατεξουσοδότηση πράξεων προβλέπει το Κοινοβούλιο εφόσον θέλει να διευκρινίσει την έννοια της εξουσιοδότησης τώρα για το 6 για την χωρητικότητα, των όγκων. Ο χρόνος κοινοποίησης όπως είπα μπορεί κάτι εξουσιοδότηση να μειωθεί Ω τώρα το μόνο κριτήριο που χρησιμοποιείται για τη μείωση είναι το τύπο του σκάφους. Σκεφτήκαμε, εγώ δηλαδή σκέφτηκα, ότι ο μικρός όγκος, η μικρή χωρητικότητα του φορτίου μπορεί να είναι και αυτό ένα κριτήριο. Και αυτό με το logbook, διότι ξέρουμε ότι όσο πιο μικρός είναι ο όγκο, τροπολογία 6 εννοώ, όσο πιο μικρό, λοιπόν είναι ο όγκο, τόσο αναλογικά μεγαλύτερη η πιθανότητα σφάλματος. Άρα μεγαλύτερη ανεκτικότητα για τους μικρούς όγκους. Εδώ έχουμε μια συζήτηση, αλλά ακούω διαφορετικές απόψεις ε, για το, τι, για το πώς βλέπουν οι συνάδελφοι την τροπολογία 10 και για τα επιστημονικά δεδομένα. Όντως, είτε θα χρησιμοποιήσουμε τον παλιό κανονισμό, είτε τον νέο θα πρέπει να είμαστε συνεπεί εδώ και απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι ανακαλύπτω ότι δεν θα υπάρξει αναθεώρηση πριν το 2015, δηλαδή κανονισμό ελέγχων. Θα προκύψει από τον παλιό βασικό κανονισμό, δεν ξέρω πώ θα γίνει αυτό στην πράξη, αλλά αυτό ακούσαμε. Και αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια διατησία μεταξύ μα. Δεν μπορούμε για το ένα άρθρο να παίρνουμε τον παλιό κανονισμό περί ελέγχων και στο άλλο άρθρο να παίρνουμε τον άλλο βασικό κανονισμό, τον καινούριο θα πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ συναδέλφων του Κοινοβουλίου αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Κοινοβούλιο για να επιλέξουμε την κατάλληλη νομική βάση. Απαντώ έτσι λοιπόν κυρία Φράγκα στην ερώτησή σας αλλά πραγματικά καλό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει υπόψη. Κατά τα καλύτερα για το τέλος, τροπολογία 13 14 δηλαδή. Για την αξιολόγηση. Με συγχωρείτε αλλά παραμένω και επιμένω στη συνθήκη. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι να ελέγχει τις καθοδότησης πράξεις. Ε, έχουμε εκχωρήσει κάποια ε, εξουσία, οπότε πρέπει εκ των υστέρων να δούμε πώς ε, αξιοποιήθηκε αυτή η ευκαιρία. Τώρα, αν δεν σας αρέσει η διατύπωση, αυτό συζητιέται, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπορεί να ασκεί την εξουσία ελέγχου που έχει το Κοινοβούλιο. Όχι όπως γίνεται σήμερα, απλώς να ανταλλάζουμε ηλεκτρονικά μηνύματα που χάνονται κάπου στους διαδρόμους τέλο πάντων πιο συγκεκριμένα στα κανάλια των ηλεκτρονικών δικτύων. Όχι, μόνο να τα συζητάμε αυτά και νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και σε κάθε περίπτωση προκειμένου να έχουμε μια συνολική αποτίμηση των κατεξοδότηση πράξεων του κανονισμού ελέγχου, αυτό μας οδηγεί σε, μια, ε, ε, σε έναν έλεγχο ανατριετία. Δεν πρόκειται για μια δυσανάλογη απέτηση σε σχέση με τις δικές μας ευθύνες να ελέγχουμε εκ των υστέρων τις οι πράξεις. Τώρα την ε, εφαρμογή μπορούμε να τη δούμε και με λεπτομέρειες αργότερα. Και για την τροπολογία 13. Δεν είναι επί της ουσίας το θέμα καθόλου και θα σας εξηγήσω γιατί. Μιλάμε για ξεκάθαρη λισαβονοποίηση εδώ. Δι, γιατί, διότι πριν τη συνθήκη της Λισαβόνας η χάρτα των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν ήταν προσαρτημένη στην ε, συνθήκη. Από νομική σκοπιά δεν οφείλαμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες της χάρτας. Από την θέση σε ισχύ της Λισαβόνας και μετά, η χάρτα έχει προστατευτεί στην συνθήκη. Είναι μέρος της συνθήκης. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε κανονισμός εγκρίνεται από εμά θα πρέπει να συνάδει με τη χάρτα. Δεν λέω λοιπόν, κύριε Πέρες, ότι ως έχει το άρθρο αντιφάσκει με τη χάρτα. Δεν το λέω έτσι. Λέω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Διότι όντως δεν συνάδει με το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνο επί του οποίου να επιβάλλεται η κύρωση. Δεν λέω ότι πρέπει να είναι αναγκαστικά ο πλειοκτήτης, Συμφωνώ με την περιγραφή που κάνατε. Την περίπτωση ο πλειοκτήτης με την πίεση που ασκεί στους ε, εργαζομένους του τελικά εκείνο να φταίει για τη λαθρέα ε, αλία ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση. Αλλά δεν είναι απαραίτητο έτσι. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε περί ευθύνης. Δεν μπορείτε να λέτε ότι κάθε φορά φταίει ο πλειοκτήτης. Ποια είναι η συνέπεια στις περιπτώσεις που δεν είναι υπεύθυνο ο πλειοκτήτης, δεν υπάρχει κανένας λόγος και αυτό είναι ε, πρωτογενές δίκαιο της συνθήκης της Λισαβόνας, δεν μπορεί να αναλαμβάνει ευθύνες που δεν είναι δικές του. Μιλάμε λοιπόν για λισαβονοποίηση με εφαρμογή των όσων προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας σε όλο το εύρος συμπεριλαμβανόμενη της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Καταλαβαίνω ότι η συζήτηση ανοίγει, αλλά μιλάμε για το φάσμα μέτρων τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Το θέμα αυτό ε, δικαίου δεν ε, είχε φυγεί ω τώρα. Εάν όμω ένα άρθρο αντιφάσκει με τη συνθήκη, ε, τι πρέπει να γίνει. Λόγω λισαβονοποίηση πρέπει να το προσαρμόσουμε. Αυτή είναι η δική μου νομική ανάγνωση των πραγμάτων θα πρέπει τουλάχιστον να ρωτήσουμε τους ε, ειδικού περί δικαίου για το θέμα αυτό. Δεν θέλω φυσικά αυτή η νομική ανάλυση να καθυστερήσει την ψήφιση της έκθεσης. Θα μπορούσε ίσως να διορθώσει εκ των υστέρων ή να, να γίνει πριν την ε, ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ξέρουμε ποια είναι τα παρασκήνια και διαδικασίε αυτού του σώματο, ξέρουμε ποιε είναι οι δυνατότητε που υπάρχουν, αλλά θεωρώ ω εισηγήτρια ότι ω προ τη λισαβονοποίηση θεωρώ αδιανόητο να μην εναρμονιστούν όλα αυτά με τη συνθήκη. Ειδικά αυτό το σημείο που αυτή τη στιγμή δεν συμφωνεί με τη συνθήκη. Απευθύνομαι λοιπόν στην νομική υπηρεσία, μάλλον στον πρόεδρο, γι' αυτό απευθύνεται αρχικά στον πρόεδρο τη Επιτροπή μα, για να μα πει τι μπορεί να γίνει. και πόσος χρόνος χρειάζεται για τη λισαβονοποίηση προκειμένου να ε, συναρμοστεί ε, το, όσα προβλέπει η Χάρτα Θεμελιδών Δικαιωμάτων και με την ίδια τη συνθήκη, εφόσον έχει προσαρτηθεί εκεί. Ευχαριστώ κύριε Θωμά. Σημειώνω αυτό που μου είπατε και θα το δούμε. Υπάρχουν άλλες ε, ερωτήσεις. Όχι. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την εξέταση αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης μέχρι τις 28 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες. Κύριε Τόμα, παρακαλώ. Ναι. Έχω ένα αίτημα παράτασης της προθεσμίας για την ε, υποβολή τροπολογιών. Ναι, ήθελα να ζητήσω μέχρι τις 28 Οκτωβρίου και τώρα συνειδητοποίησα ότι αυτό μόλις τώρα είπατε. Ναι, ναι, ήδη το έχω εγκρινεί. Τροπολογή λοιπόν μέχρι 28 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης σε σχέση με το Μαγιότ ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό πάμε τώρα. Η έκθεση αυτή είχε ανατεθεί στην ΚΟΕ τον Ιούλιο. Ο Ζωάο Φερέιρα είναι ο εισηγητής. Σήμερα λοιπόν θα μας κάνει μια παρουσίαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ από την Επιτροπή για το θέμα της Μαγιότ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε αυτή την πρόταση. Γιατί? Διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε η Μαγιότ να θεωρηθεί αξόχως ε, απόκεντρη περιφέρεια από την 1η Πρώτου του 2014. Βάσει της απόφασης αυτής, λοιπόν, η Γαλλία μας υπέβαλε αίτημα σύνταξης γνωμοδότησης, δηλαδή ποια μέτρα δεν είναι σε θέση να τηρήσει και με ποια μέτρα δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί η Μαγιότ. Και το συμπέρασμα πράγματι ήταν ότι η Μαγιότ δεν είναι καθόλου έτοιμη να προσαρμοστεί στο κεκτημένο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και ότι δεν θα προλάβει να το κάνει μέχρι την 1η Πρώτου του 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε λοιπόν να γίνουν κάποιες προσαρμογές στην κοινή αλληλευτική πολιτική για να μπορέσει η Μαγιώτα να ενσωματωθεί σταδιακά και να αφομοιώσει σταδιακά το κεκτημένο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στο αίτημα της Γαλλίας αλλά επίσης τεκμηριώνεται λόγω της γνώσης που έχουμε περί της κατάστασης στην Μαγιώτα. Και πολύ απλά λοιπόν, με απλά λόγια, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγκυται στο εξής. Παρουσιάζουμε ορισμένα βασικά στοιχεία της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και πιο συγκεκριμένα τα εξής. Το αρχείο, το μητρό για τους αλλιευτικούς τόλους, τις συνθήκες για την ετικετοθεσία της σήμανση και ε, τον κανονισμό για τους ελέγχους. Αξιοποίησε την ευκαιρία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει και κάποιε τροποποιήσει σε όλα αυτά τα κείμενα, τα οποία, τις οποίες θεωρεί απαραίτητε ούτως ή άλλως. Όχι μόνο γιατί η αλλω οχι μονο γιατι η μαγιωτε δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην κοινιαλιευτική πολιτική, αλλά ούτω ή άλλω πρέπει να επέλθουν αυτέ οι τροποποίησει για καλύτερη ενοποίηση και ολοκλήρωση στην πολιτική αυτή. Και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στην παράταση, στην επέκταση στα 10 μίλια της ζώνης αποκλειστικής ε, δραστηριότητας στη Μαγιώτα. Αυτό ισχύει και για τη Μαδέρα και για τις Αζόρες νήσους ούτως ή άλλως. Ε, είναι λογικό να ισχύσει και για τη Μαγιώτα. Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, αυτή η αποκλειστική ε, πρόσβαση μέχρι τα 10 μίλια πρόσβαση της Μαγιότ κατά πάσα πιθανότητα ε, ε, ισχύει και θα ισχύσει και για τις άλλες εξόχως από κέντρες περιφέρειες. Να σας πω και να σας περιγράψω συντομία πώς έχει η κατάσταση στη Μαγιώτα από πλευράς αλλιευτικής δραστηριότητας. Είναι ένα ηφαιστικό νησί που περιβάλλεται από κοραλιογενή ύφαλο. Μεταξύ του κοραλιογενούς υφάλου και του ηφαιστιακού νησιού έχουμε αυτή την λιμνοθάλασσα με όχι πολύ βαθιά ύδατα, ενώ ο κοραλιογενής ύφαλος είναι αρκετά μακριά από την ακτή. Είναι μία από τις μεγαλύτερες λιμνοθάλασσες ε, με κορεαλιογενείς υφάλους στον κόσμο. Αυτά για τη γεωμορφολογία της περιοχής. Μέσα Εκεί λοιπόν έχουμε ηχθιαποθέματα εξαιρετικά ευαίσθητα στα οποία γίνεται υπερεκμετάλλευση. Παραδοσιακά οι ντόπιοι αλίευαν, ψάρευαν εκεί και ε, τώρα υπάρχει ε, υπερεκμετάλλευση στα ηχθιαποθέματα που είναι ανάμεσα στα ρηχά νερά της λιμνοθάλασσης, λιμνοθάλασσας. Έξω από τον κοραλιογενή ύφαλο έχουμε πολύ βαθιά ύδατα και είναι σημείο από το οποίο περνούν τα μεταναστευτικά είδη. Τώρα, ο αλευτικός θόλος της Μαγιώτα αποτελείται από τρεις βασικούς ε, τομείς. Έχουμε μεγάλα αλλιευτικά σκάφη ε, που ψαρεύουν τόνο, κυρίως και όλα αυτά τα τονοειδή έχουν σημαία γαλλική ή άλλη. Δεν ξεκινούν από τη Μαγιότ, αλλά ξεκινούν από το νησί της Ρεουνιών και είναι ε, δραστήρια αυτά τα λευτικά σκάφη σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε και άλλο στόλο που είναι τα μικρά σκάφη με παραγάδια και δίχτυα, πολύ μικρά λιευτικά σκάφη, μηχανοκίνητα και αλλιεύουν τα μεγάλα ε, ψάρια που μεταναστεύουν, δηλαδή τσιπούρες, ξυφίες, ε, μεγάλα τονοειδή και το καθεξής. Και τέλος, ε, έχουμε τις, τα σκάφη Yamaha. Τα έχουν ονομάσει έτσι γιατί είχαν εξολέμβιο κινητήρα Yamaha. Είναι κάτι που είχε ε, προωθήσει η ΦΑΟ σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, να, να τέτοια, τέτοιου είδους μικρά φουσκωτά ή σκάφη, αν θέλετε, με εξολέμβια μηχανή κινητήρα. Αλλά είναι επικίνδυνα. Είναι ασταθή. Είναι ασταθή η λέμβη αυτή. Δεν είναι πολύ αποτελεσματική. Είναι επικίνδυνες και η αλευτική τους δυνατότητα ε, είναι περιορισμένη. Είναι αν, ανοργάνωτη, αν θέλετε, αυτού του είδους η ελευτική δραστηριότητα. Δεν ε, εκφορτώνουν σε συγκεκριμένες ηχθιόσκολες. Δεν υπάρχει αλυσίδα εμπορίας και διάθεση στην αγορά η οποία μπορεί, να μπορεί να εντοπιστεί και να παρακολουθηθεί. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι πολύ υπανάπτυκτη η δραστηριότητα αυτή δεν είναι καν υπό ανάπτυξη γιατί πολύ πρόσφατα κάναμε απογραφή ε, του πληθυσμού των αποθεμάτων πολύ πρόσφατα θεσπίσαμε δηλαδή ε, μηχανισμούς παρακολούθησης έχουμε μεγάλο αριθμό λαθρομετανάστευσης και πάρα πολλές ε, τέτοιες βάρκες χρησιμοποιούνται άναρχα και δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Δεν υπάρχει ένας μόνος ιδιοκτήτης, μια ολόκληρη οικογένεια μπορεί να έχει μια, μια τέτοια βάρκα. Είναι δηλαδή κλάδος, είναι μέσο πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Υπ' αυτή την έννοια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το κομμάτι του αλλιευτικού της στόλου, της Μαγιότ, που είναι το πιο δύσκολο να συμμορφωθεί με την κοινή αλλιευτική πολιτική, είναι αυτό το τρίτο κομμάτι των, με τις βάρκες τύπου Γιαμάχα και έχουμε και τις πυρόγες που είναι μικρές βάρκες, αυτοσχέδιες που έχουν ε, ε, φτιαχτεί από τον κορμό ενός δένδρου και εκεί βεβαίως οι άνθρωποι αλλιεύουν για εσωτερική, προσωπική, οικογενειακή κατανάλωση και σπανιότατα ε, πολλούν τα, ό,τι τους έχει περισσέψει στην άκρη του δρόμου, στον αυτοκινητόδρομο ή σε αυτοσχέδια παραπήγματα. Δεν είναι λοιπόν εμπορική αυτή η δραστηριότητα κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άρα δεν εντάσσεται στην κοινή αλληλευτική πολιτική και αυτές οι πυρόγες δεν μπορούν να θεωρηθούν αλληλευτικά σκάφη. Μπορεί αργότερα να θεωρηθούν ως τέτοια, αλλά όχι προς το παρόν, κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές οι οι πυρόγες που είναι φτιαγμένες από κορμό δένδρου κατατάσσονται σε αυτό το οποίο στην Ευρώπη ονομάζουμε μη επαγγελματική αλληλεία. Θα ήθελα να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι εμείς ε, μιλούμε για την καταχώρηση του στόλου και το μητρό του στόλου. Έχουμε λοιπόν ε, τα σκάφη τύπου Yamaha που θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν σε αυτό το μητρό, όχι άμεσα και όχι απαραίτητος και όχι με πλήρη συμμόρφωση όλων των προϋποθέσεων των κοινοτικών. Να ενταχθούν στο μητρό σταδιακά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Εν τω μεταξύ όμως, από σήμερα μέχρι ε, τα τέλη του 2016, για να μην θεωρηθεί αυτό αυτή η βάρκα τύπου Yamaha ως βάρκα η οποία ασκεί λαθρέα, άναρχη και παράνομη αλία. Να κάνει η Γαλλία προτείνουμε μια προσωρινή καταγραφή για να εντοπίσουμε τους ιδιοκτήτες και να μπορούμε να έχουμε έναν ελάχιστο έλεγχο μέχρι να συμμορφωθούν πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τώρα, ως προς την πρόσβαση στην αλληλευτική δραστηριότητα μέχρι τα 10 μίλια στα χωρικά ύδατα της Μαγιόντ η επέκταση αυτή μέχρι τα 10 μίλια δεν είναι κάτι που προτείνουμε ε, γιατί ε, δεν μπορούν αλλιώς να αλλιεύσουν, αλλά γιατί το θεωρούμε απαραίτητο προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση γενικότερη, να υπάρχει ευθυγράμμιση και σε σχέση με άλλα νησιά. Για την καλύτερη προστασία των αποθεμάτων, για να αποφύγουμε οι μεγάλες ε, τα μεγάλα αλλιευτικά σκάφη από άλλες χώρες και τα μεγάλα αλλιευτικά σκάφη ε, της Μαγιώτε να αλλιεύσουν στις ίδιες περιφέρειες και τις ίδιες περιοχές με τις βάρκες τύπου Yamaha προτείνουμε να επιτρέψουμε στις βάρκες τύπου Yamaha να έχουν αλλιευτική δραστηριότητα μέχρι ε, στα 25 μίλια. Τώρα, ως προς τα πρότυπα ετικετοθεσίας, η Επιτροπή προτείνει παρέκκληση μόνο πάλι για αυτό το 1 τρίτο του κλάδου, για το κομμάτι του κλάδου που έχει να κάνει με τις βάρκες Yamaha, τύπου Yamaha, διότι δεν υπάρχουν τα ε, κατάλληλα ε, κανάλια επικοινωνίας και ε, Διάθεση στην αγορά. Θεωρούμε ότι προς το παρόν δεν είναι απαραίτητο αυτές οι βάρκες τύπου Yamaha να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις σε θέματα ετικετοθεσίας και σήμανσης. Και ως προς τον κανονισμό ελέγχου η Επιτροπή προτείνει παρέκκληση μόνο επί των άρθρων όπου υπάρχουν πραγματικές δυσκολίες που ζητούν να ε, επισημανθούν τα αλλιευτικά εργαλεία, τα αλλιεύματα και καθεξής. Ο κλάδος δεν είναι σε θέση να τα εφαρμόσει όλα αυτά, δεν έχει οριμάσει αρκετά για να μπορέσει να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίω, όπως και με το Μητρό του Αλευτικού Στόλου, και εδώ η Επιτροπή προτείνει η Γαλλία να είναι αυτή που ε, να θεσπίσει ένα προσωρινό ε, καθεστώ ελέγχου με κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις, έτσι ώστε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη πρώτη του 2014, η αλία γύρω από αυτά τα νησιά στην πολύ κοντινή ε, περίμετρο αυτών των νησιών να είναι βέβαια η αλληλεία από τις βάρκες τύπου Yamaha, αλλά να μην θεωρηθεί και να μην μπορεί να θεωρείται λαθρέα, άναρχη και παράνομη αλληλεία. Ζητούμε από τη Γαλλία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014 να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης, διασφαλίζοντας ότι αυτό το σύστημα ελέγχου ε, σιγά σιγά θα αφομοιωθεί και θα ενσωματωθεί από τον κλάδο, από την ε, αγορά και από τα αλληλευτικά σκάφη. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έκανε την παρουσίασή της. Την βρήκα διεξοδική. Ακούσαμε και για την πρόταση κανονισμού και για το τι διακυβεύεται. Στόχος του κανονισμού είναι να αλλάξει μια σειρά κανόνων και κανονισμών το χώρο της αλίας για να μπορέσουμε να καλύψουμε και την Μαγιότ που άλλαξε πρόσφατα καθεστώς μετά την απόφαση του Συμβουλίου του 2012. Πάβει να είναι υπερπόντιο έδαφος και γίνεται εξόχως από κεντρή περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα αρχίζει να ισχύει η, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τομέα της αλίας, στη Μαγιότ, κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει μια σειρά από κανόνες δεδομένου της ιδιαίτερης κατάστασης αυτής της εξόχως απόκεντρης περιοχής. Έτσι μάλιστα όπως μας την παρουσίασε η Επιτροπή ένα κανονισμός τεχνικών μέτρων, κανονισμός κοινή οργάνωση αγοράς που ισχύει ε, ήδη ο κανονισμός ελέγχων, ο κανονισμός για την έρευνα και την ε, βιώσιμη αξιοποίηση των, ε, των πόρων και ούτω καθεξής. Νομίζω η προσαρμογή αυτή, η συμπερίληψη της Μαγιότ στο κοινοτικό σύστημα θα πρέπει να γίνει με τρεις βασικές μέρημνες υπόψη μας. Νομίζω τις ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά πρώτον, έχοντας υπόψη τις ιδιαίτερα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Μαγιότ, με το πολύ ιδιαίτερο στάδιο ανάπτυξης του αλληλευτικού του τομέα, το, πολύ, το, το ιδιαίτερο χαρακτήρα των ε, αλληλευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνται εκεί, τα οποία είναι διασκορπισμένα σε όλο το νησί, χωρί συγκεκριμένα σημεία πρόσδεση, χωρί ε, συγκεκριμένο εξοπλισμό. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε χρόνο στη Μαγιότ για να προσαρμοστεί στην νομοθεσία μα. Αυτό είναι η πρώτη μέρημνα. Η δεύτερη, κάτι που ανέφερε ούτω ή άλλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να αναγνωρίσουμε τις ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων που απαντά κανένας στη Δηλαδή, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οικοσυστήματα πλούσια από την άποψη της βιοπικιλότητας, με ιδιαιτερότητες που ακούσαμε, με την παρουσία κορυλιαγενούς ε, υφάλου, το οποίος καθορίζει μια λιμνοθάλασσα με νερά ενώ από την άλλη υπάρχουν τα είδη που βρίσκονται γύρω από τον και ύφαλο με άλλα χαρακτηριστικά, αυτή, αυτός ο πλούτος, αυτή η επικοινότητα θα δικαιολογούσε και δικαιολόγησε τη δημιουργία του φυσικού πάρκου της ε, Μαγιότ. Το ότι δεν είναι κατάλληλη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ιδιαιτερότητες της Μαγιότ είναι κάτι που δεν θα πρέπει να μας κάνει να πάψουμε να προστατεύουμε αυτές τις ε, αξίες της φύσης και τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος εκεί. Και κάτι ακόμη, το τρίτο στοιχείο. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γίνουν επιλογές και μάλιστα έχοντας υπόψη το στόχο προστασίας των φυσικών αποθεμάτων του, της νήσου. Ε, επιλογές από την άποψη της διαχείρισης. Ναι, αλλά πρώτα απ' όλα πρόσβαση να υπάρχει για το στόλο του νησιού. Ε, το, τα μικρά αυτά σκάφη, τα αυτοσχέδια σκάφη στους ελευτικούς πόρους και μετά για τα μεγαλύτερα σκάφη. Για τα μεγάλα αθηναλιευτικά λόγου χάρη τα οποία θα πρέπει να αλλιεύουν όχι στη Μαγιότ μέσα αλλά σε άλλα μέρη. Αυτές είναι οι τρεις βασικές ε, μεταβολές. Νομίζω καλύπτονται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά περιθώριο για λίγες προσαρμογές ακόμη υπάρχει. Ε, είτε για την πρώτη από τις μερίμνες που ανέφερα, δηλαδή το χρόνο που μπορούμε να δώσουμε στη Μαγιότ για να ολοκληρώσει το μητρό αλληλευτικών σκαφών, τέλος πάντων το νεολόγιο, για να μπορέσει να ενταχθεί στην κοινή οργάνωση αγοράς, να προβλέψει τα ιδιαίτερα μέτρα που χρειάζονται για την ε, ε, προστασία των ηχθιαποθυμάτων της νήσου. 24.000 είπαμε στη μία περίπτωση, 20.000 ε, στην άλλη. Καλύτερη αντιστοιχία πρέπει να βρεθεί με την περιοχή του φουσικού πάρκου της Μαγιώτη πρέπει να δούμε ποιες είναι ακριβώς οι αξίες της φύσης που θέλουμε να... και οι τιμές που θέλουμε να προστατευτούν. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική συλλογιστική όταν μιλάμε για συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Άλλη θα είναι συλλογιστικοί για το φυσικό πάρκο και άλλη για τις υπόλοιπες περιοχές. Τα 24 ή τα 6 μίλια είναι διαφορετικά, θα πρέπει να ισχύουν διαφορετικά εάν μιλάμε για το φυσικό πάρκο ή όχι. Έτσι κι το φυσικό πάρκο της Μαγιότ ε, εντοπίστηκε με, την, ε, με, κριτήριο το να προστατευτούν οι φυσικές τιμές που θέλαμε να προβλέψουμε και όχι με βάση τα 6 τα 24 μίλια. Αυτό θα πρέπει να είναι το κριτήριο που θα μας καθοδηγήσει. Οι αλλαγές αυτές, οι προσαρμογές πιστεύω μπορούν να γίνουν ε, καλύπτοντας μας ακόμα περισσότερο ως προς αυτές τις τρεις μέρημνες. Τα είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να εγκριθούν, απλώς λίγο περισσότερο να ενισχυθούν. Δεν έχω άλλες προτροπές να κάνω, μπορώ να κλείσω εδώ. Ευχαριστώ κύριε Φράγα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή και τον εισηγητή. Με εντυπωσίασε η κατάσταση του αλληλευτικού τομέα στη Μαγιότ γιατί ιδίω ένα τμήμα όπως το περιγράφει είναι αξιοσημείωτο. Αυτές οι υπερπόντιες περιοχές δεν ε, ε, προσπάθησαν τα κράτη στα οποία ανήκουν να του επιβάλλουν κάποιε υποχρεώσει. Δεν υπάρχει ούτε νεολόγιο. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα για τα 100 μίλια. Αυτό που εξηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι θέλουν να εξισώσουν την κατάσταση με τις τρεις άλλες υπερπόντες περιοχές που είναι μία Ισπανική και δύο Πορτογαλικές. Εντάξει. Αλλά θα ήθελα και περισσότερες εξηγήσει γιατί πρέπει να υπάρχει απόλυτη ισοτιμία στην αντιμετώπιση όλων των υπερποντίων περιφερειών. Όταν έγινε η εξαίρεση των 100 μιλίων για τα Κανάρια, τη Μαδέρα και τις Αθόρες, ήταν πολιτική συμφωνία. Κατά την ένταξη της Ισπανίας και την Πορτογαλία. Ήταν πολιτική συμφωνία. Δεν έχει καμία επιστημονική ή άλλη βάση. Θα ήθελα να μάθω εάν για την περίπτωση της Μαγιώτη υπάρχει επιστημονική βάση. Γιατί αν δεν υπάρχει, ε, τώρα το ότι είχε υπάρξει μια πολιτική συμφωνία, αυτό είναι άλλο, δεν σημαίνει πως πρέπει να εφαρμόζεται παντού. Δεν θα πω άλλα, αλλά θα ήθελα να μάθω αν είναι φυσιολογική αυτή η διαδικασία. Δεν θα έπρεπε να έχει κάνει κάτι η Γαλλία προηγουμένω. Και να μου πείτε λίγο περισσότερα για αυτό το σχέδιο αύξησης ε, της ε, χωρητικότητας του στόχου στον Ινδικό. Διότι εάν δεν σεβαστούμε ούτε χώρο, ούτε χωρητικότητα, θα ήθελα να μου εξηγήσει τι είναι αυτό το σχέδιο. Κατά πόσο θα ευξηθεί η χωρητικότητα του στόλου, πώς θα τα λύσουμε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Φράγα. Θα μιλήσω από πλευράς του κυρίου Καντέκ που μου ζήτησε να διαβάσω ένα έγγραφο και θα το διαβάσω. Είναι τα λόγια του κυρίου Καβέκ τα οποία διαβάζω. Την 1η Πρώτου 14 το Μαγιότ ε, θα γίνει υπερπεριφερειακή περιοχή. Με βάση το άρθρο 349 της ε, Συνθήκης της Ένωσης, καλό αυτό για τη Μαγιότ, που θα ήθελε να λάβει τις ιδιαιτερότητές της ε, η Ένωση. Είναι πολύ απομακρυσμένη, μικρό νησί με κλίμα και τοπογραφία πολύ διαφορετικά και δυσχερή. Δεν είναι εύκολο να εφαρμόσει από την 1η 1η 14 στον τομέα της αλληλείας το κοινωνικό δίκαιο. Χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστεί η Μαγιώτα στους νέους κανονισμούς Πάντα χρειάζεται χρόνος προσαρμογής για την ε, συμμόρφωση στις ε, ενωσιακές ρυθμίσεις. Πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποιες εξαιρέσεις για ένα κάποιο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, χρόνος προσαρμογής στη σήμανση που προβλέπει το άρθρο 42 της κοινή οργάνωσης αγοράς, διότι η αγορά στη Μαγιότ είναι κατακαιρματισμένη, υπανάπτυκτη. Ε, επίσης, ε, χρόνο για να εγγραφούν στον ιολόγιο, γιατί υπάρχουν διάφορα σκάφη κάτω από 10 μέτρα που δεν έχουν ε, τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και περιορισμός ε, για κάποια είδη μόνο για, αλήψεις για κάποια είδη μόνο για τα σκάφη που, είναι, ε, που εκφορτώνουν στη Μαγιότ με βάση το άρθρο 34α που περιορίζει δραστηριότητες στα 24 μίλια για να επιτρέψουμε να τους προστατεύσουμε από τη βιομηχανική τον αλίευση που θα τους αφαιρούσε θηναλευτικού πόρους. Θεωρούμε ότι πρέπει να διατηρηθεί η κανονική ε, νομοθετική διαδικασία που πρότεινε η Κομισιόν το 43-2. και με βάση το άρθρο 49 πρέπει να ε, ε, προσθεθεί και το άρθρο 49 γιατί αυτό ρυθμίζει πώς εφαρμόζεται το κοινωνικό δίκαιο στις άκρος περιφερειακές περιοχές. Αυτή είναι η θέση του κυρίου Καντέκ. Εφόσον δεν μου ζήτησε άλλο το λόγο, η Κομισιόν απαντήσει δύο ερωτήσεις που τέθηκαν για τα 100 μίλια και την αύξηση του, της ε, χωρητικότητας. Ευχαριστώ. Να απαντήσω και σε μια τρίτη που νομίζω είναι η πρώτη που έκανε η κυρία Φράγα για τις υποχρεώσεις των ε, υπερποντίων περιοχών. Ε, ε, φυσικά δεν είναι υποχρεωμένε, αλλά μπορούν να το κάνουν ε, ε, εθελουσίω. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένε να τηρούν το κοινοτικό δίκαιο. γιατί τη βάση των 100 μιλίων και αν έχουμε επιστημονική ε, θεμελίωση. Υπάρχουν μια σειρά και επιστημονικά αλλά και πολιτικά επιχειρήματα και status quo επιχειρήματα. Διότι, κοιτάξτε, υπάρχει αυτή, αυτός ο περιορισμός. Από την 1η πρώτου 14 το ότι θα εφαρμοστεί κάτι διαφορετικό δεν αλλάζει την κατάσταση. Άρα θέλουμε να διατηρήσουμε το status quo επιστημονικά, σίγουρα. Υπάρχει πολλής τόνος και συναφή ε, δηλαδή ιδιαίτερα αποδημητικά ε, είδη, κοντά. Είναι ένα ιδιαίτερο είδος ε, αλίευσης, αλίας, και είναι ιδιαίτερα ευάλωτη η πόρη. Να περιορίσουμε την πρόσβαση στα σκάφη που έρχονται από μακριά, που έχουν περισσότερες δυνατότητες αλίευσης από τους ε, ντόπιου με κατά κάποιο τρόπο διατηρεί τα αποθέματα. Υπάρχει το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό θέμα γενικότερα. Θα διαπιστώσετε ότι στις ιδεολογικές σκέψεις σχεδόν αντιγράφουμε την ιδεολόγηση που είχε τεθεί στην περίπτωση των Αζωρών, της Μαδέιρα και των Καναρίων. Ποια είναι τώρα τα σχέδια ανάπτυξη τη επιτροπή για τον τόνο στον Ινδικό. Νομίζω ότι το 2005 λήφθηκε η απόφαση να παγώσει η χωρητικότητα, η δυνατότητα λίευσης μάλλον των σκαφών. Τώρα με την ε, αποτίμηση της ε, κατάστασης των αποθεμάτων είχαν μελετήσει τους ξηφίες συγκεκριμένα Προτείνεται τώρα λοιπόν μια απόφαση που θα ήθελε να παγώσουν οι στόλοι, να μην αυξηθεί η χωρητικότητά τους, η δυναμικότητά τους, ε, με βάση την κατάσταση μιας συγκεκριμένης χρονιάς που δεν θυμάμαι ποια είναι. Αλλά παράλληλα προβλέθηκε και μια εξαίρεση σε αυτήν την απόφαση που θα επέτρεπε στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά να αυξάνουν τους στόχους τους για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Για να το κάνουν αυτό έπρεπε να υποβάλουν σχέδια ανάπτυξης στην Επιτροπή Ινδικού. Υποβλήθηκαν αυτά τα σχέδια το ένα μετά το άλλο και στην περίπτωση της Μαγιώτ η Γαλλία εκ μέρους της Μαγιώτ υπέβαλε το τελευταίο σχέδιο ανάπτυξης το 2011. Και η Επιτροπή του Ινδικού το εξέτασε και κανένας ούτε η Ένωση δεν υπέβαλε αντιρρήσεις. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι καταρχήν, μόνο καταρχήν, θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε αυτή την αύξηση του δυναμικού του στόλου της Μαγιότ στο μέλλον με βάση τα σχέδια ανάπτυξης. Βέβαια, επειδή τα μεγάλα Αθήνα αλλιευτικά έχουν τεράστια δυνατότητα αλλιεύσης δυσανάλογα μεγαλύτερη από τα άλλα δύο τμήματα του στόλου η Κομισιόν θεώρησε ότι θα ήταν πιο λογικό με την κοινοτική προσέγγιση στην Επιτροπή του Ειδικού να διατηρηθούν τα αποθέματα, να μην αυξάνεται το δυναμικό. Θα ήταν λοιπόν πιο λογικό να μην αυξηθεί αυτό το τμήμα του στόλου που είναι αυτό που έχει τις περισσότερες δυνατότητες. Υπάρχουν πέντε μεγάλα γρηγροί και όταν ε, λέω μεγάλα εννοώ μεγάλα, πάνω από 80 μέτρα που ήδη λειτουργούν υπό σημαία Και το σχέδιο ανάπτυξης προέβλεπε άλλο ένα η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτό θα ήταν αύξηση 20% και ότι αυτό δεν είναι συμβατό με την προσέγγιση της Ένωσης στην Επιτροπή Ινδικού. Η αύξηση για τα άλλα δύο τμήματα είναι επίσης ε, σημαντική. Συνολικά όμως τα άλλα δύο τμήματα έχουν πολύ μικρότερες δυνατότητες από ότι τα θυναλευτικά, τα παραγαδιάρικα λοιπόν. Αυτοί οι άλλοι τομείς λοιπόν συμβάλλουν και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αλληλείας στην Ίσο. Τέλος, για τα σκάφη μάχα Το σχέδιο ανάπτυξης προέβλεπε ένα ανώτατο όριο που στην ουσία δεν αυξάνει το δυναμικό. Απλώς ε, κατοχυρώνει το υπάρχον δυναμικό. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι να εξχρονιστούν, να είναι πιο ασφαλή αυτά τα σκάφη, να πληρούν καλύτερα τις συνθήκες υγιεινής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φράγα. Ευχαριστώ. Ένα θέμα μόνο θέλω να σχολιάσω που είπατε και δεν το καταλαβαίνω και πολύ καλά. Πράγματι, η ζώνη των 100 μιλίων θα είχε νόημα για την προστασία των ειδών μόνο αν μιλούμε για εξόχως μεταναστευτικά ή αποδημητικά είδη. Αλλά δεν, δεν καταλαβαίνω το επιχείρημά σας. Ο κύριος Φερέιρα για την ε, τελική απάντηση στη συζήτηση. Η δημιουργία ζωνών 6 μιλίων σκοπό έχουν από τη μια να προστατεύσουν τους πόρους αλλά από την άλλη και τους τοπικούς στόλους. Αυτός ο διτός στόχος επιδιώκεται ακριβώς με αυτή την παρέκκληση. Από τη δική μου την οπτική γωνία οι στόχοι αυτής της παρέκκλησης επιτυγχάνονται με καλύτερο τρόπο και το ίδιο κάναμε λόγω χάρη για τις Ασόρες και τη Μαδέρα εάν αντί για 6 μίλια βελτιώναμε την αντιστοιχία με την πραγματική παρουσία των φυσικών πόρων όπως απαντώνται στο συγκεκριμένο σημείο και στις Ασόρες και στη Μαδέρα αλλά και στη Μαγιότ υπάρχουν σημαντικά είδη που πρέπει να προστατευθούν είτε για την ε, αυτή, ε, αυταπόδεικτη αξία τους είτε για τη σημασία που έχουν ε, για τους τοπικούς στόλους. Είναι εκτός όμως της ζώνης των 6 μιλίων. Αντί λοιπόν για 6 μίλια μπορεί να μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε την περιοχή αυτή με τα πραγματικά όρια του φυσικού πάρκου της Μαγιότ. Τα όρια αυτά ορίστηκαν βάσει της ανάγκης προστασίας συγκεκριμένων ε, ειδών και φυσικών τιμών που απαντώνται εκεί. Τα είπα αυτά και προηγουμένως. Και μία μόνο πτυχή που προηγουμένως την ε, παρέβλεψα. Προφανώς έχουμε να κάνουμε εδώ με προσαρμογές της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιδιαίτερη κατάσταση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας εξόχως απόκεντρης περιοχής. Βλέπουμε ότι χρειάζονται παρεκκλήσεις δεδομένου του χαρακτήρα αυτής της απόκεντρης περιοχής της Μαγιότ. Χωρίς λοιπόν να αμφισβητούμε την νομική βάση, όπως έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα τα άρθρα 43, 2 και 4... Τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λογικό μου φαίνεται να ε, καλύπτεται και το άρθρο που έχει να κάνει με τις εξόχους απόκεντρες περιοχές. Όχι να αντικαταστήσουμε ή να αλλάξουμε κάτι από αυτά που υπάρχουν, απλώς να προσθεθεί το 349 για τις εξόχους απόκεντρες περιοχές, εφόσον κατάφορα έχουμε να κάνουμε με την πρόβλεψη εξαιρέσεων, παρεκκλήσεων, ιδιαίτερων συνθήκων της Γενικής Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή. Υπ' αυτήν την έννοια, λογικό μου φαίνεται να προσθέσουμε το 349, το 349. Αφού το ή άλλως η η ε, υπάρχει στο, στο κείμενο, δεν θα αλλάξουμε κάτι, απλώς θα συμπληρώσουμε. Ευχαριστώ. Κατ' εξαίρεση θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, εν συντομία, γνωρίζετε όλοι ποια είναι η θέση της Κομισιόν για το 349. Θέλω να σημειώσω το εξής. Το 349 προβλέπεται μόνο για παρεκκλήσεις από τη συνθήκη. Έτσι το ερμηνεύει η Κομισιόν. Αλλά για αυτή την περίπτωση συγκεκριμένα από τη στιγμή που καθορίζονται, ή μάλλον να το ξαναπώ, ε, στην περίπτωση αυτή αν θεωρήσουμε τις άλλες ε, εξόχως απόκεντρες υπερπόντιες περιφέρειες, αν τις εξετάσουμε, δεν χρειάζονται τέτοια παρέκκληση ή άλλες. Βεβαίως υπόκειται στις ειδικέ περιστάσεις του ότι είναι πολύ απομακρυσμένες, έχουν ισιωτικό χαρακτήρα και το καθεξής. Η Μαγιότ χρειάζεται παρέκκληση, όχι γιατί είναι πολύ μακριά, γιατί είναι νησί, είναι απομανωμένη ή έχει γεωγραφικές ή ε, γεωμορφολογικές, κλιματολογικές συνθήκες ε, ε, δυσχερείς που τη δυσχεραίνουν. Χρειάζεται παρέκκληση λόγω επίπεδου ανάπτυξης, το οποίο είναι χαμηλό. Χρειάζεται να δοθεί χρόνος δηλαδή. Και ελπίζουμε ότι αυτές οι παρεκκλήσεις θα πάψουν να ισχύουν με... μετά από κάποια χρόνια. Και γι' αυτό δεν βασιστήκαμε στο 349. Επιμένω λοιπόν, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αρμόζει να βασιστεί κανείς στο άρθρο 349. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Λοιπόν, αρκετά με αυτό το θέμα, το συζητήσαμε πισταμένος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε απέχει από την χρήση του 349 χωρίς να προβάλλει ισχυρά επιχειρήματα. Εγώ προέρχομαι από μια πολύ απομακρυσμένη και νησιωτική περιοχή και το 349 είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει προσωπικό είναι αυτό το σχόλιο και ήθελα να το ξέρετε. Περνούμε στο σημείο 10 λοιπόν της ημερήσιας διάταξης. που είναι το 11 όπως γνωρίζετε γιατί το 11 έχει πάρει τη θέση του 10. ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν σε σχέση με την Ισλανδία και τις νήσους Φερόε. Δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσει. Ξέρετε ότι η Κομισιόν είχε συμφωνήσει να εμφανιστεί η ίδια η Επίτροπος για να εξηγήσει την κατάσταση. Από τη στιγμή που η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με την ημερομηνία Συμβουλίου Υπουργών δεν ήταν δυνατόν να έρθει η ίδια η Επίτροπος. Έχουμε πρόσωπό της η οποία θα μας εξηγήσει λοιπόν πώς έχει η κατάσταση. Είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερο στη δική μας Επιτροπή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε διότι δίνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να σας ενημερώσει για τις εξελίξεις για ένα θέμα που είναι αρκετά περίπλοκο. Και επειδή είναι τόσο περίπλοκο θα διαιρέσω την παρουσίασή μου σε τρία ε, βασικά μέρη. Πρώτον, το ιστορικό. Πώς καταλήξαμε ε, να υιοθετήσουμε αυτά τα εμπορικά μέτρα σε σχέση με τις νήσους Φερόε. Δεύτερον, πώς έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή στις διαβουλεύσεις με ε, αυτά τα νησιά για τα επόμενα χρόνια και τρίτον η διαδικασία διαιτησίας που έχει ε, ξεκινήσει εξαιτία της ε, διαμάχης μας με τις νήσους Φερόες. Τα εμπορικά μέτρα λοιπόν πώς ξεκίνησαν. Να σας υπενθυμίσω τα εξής επιγραμματικά. Το απόθεμα... Ε, ρέγκας είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Μιλούμε για ένα εκατομμύριο τόνους ετησίως και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας. Ε, ψάρια πάρα πολύ μεγάλα, με πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος και πολύ μεγάλη κατά συνέπεια εμπορική αξία. Τα διαχειρίζονται λοιπόν τα αποθέματα αυτά πέντε ε, παράκτια κράτη βάσει συμφωνίας που έχουν μεταξύ τους. Γίνεται συμβουλευτική διαδικασία μεταξύ ημών και ημών των διαφόρων των πέντε. Και όλα αυτά λοιπόν λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο ενός arrangement, μιας διευθέτησης η οποία εγκρίθηκε το 2007. Το 2007 λοιπόν έχουμε την τελευταία συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι μια συμφωνία που έχει εξελιχθεί με την πάραδο των ετών μέχρι την τελική τελευταία που ήταν το 2007. Λοιπόν, έχουμε τα ανώτατα επιτρεπόμενα αλλιεύματα βάσει συγκεκριμένου προγράμματος και έχουμε και συγκεκριμένο πρόγραμμα για την κατανομή αυτών των μέγιστων επιτρεπόμενων αλλιευμάτων και οι, νήσες, Φερόε βάσει της κατανομής μπορούν να αλλιεύσουν το 5,17% του συνολικού μέγιστου επιτρεπόμενου αλλιεύματος. Τον Οκτώβριο του 2011 οι νήσοι Φερόε ανακοίνωσαν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένες με το 5,17% με τη δική τους ποσόστοση και γι' αυτό ζήτησαν να ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη συζήτηση ε, της ποσόστοσης αυτής. Κανείς δεν αρνήθηκε να το συζητήσει και μάλιστα συμφωνήθηκαν να ε, υπάρξει μια ε, να υπάρξει ένα επιστημονικό συμβούλιο το οποίο θα έρθει σε επαφή με το Διεθνές Συμβούλιο για την Αξιοποίηση και Εκμετάλλευση των Θαλάσσιων Πόρων, ούτως ώστε να ε, υπάρξει πόρισμα για καλύτερη κατανομή των αποθεμάτων ρέγκας. Το 2011 οι νήσοι Φερόε δέχθηκαν λοιπόν να συνεχίσουν με το 5,17% και το είχαν αποδεχτεί σαν μέγιστη ποσόστοση. Τον Οκτώβριο τώρα του 2012 ξεκίνησε η συζήτηση για τα μέτρα για το 2013 και οι νήσοι Φερόε υπενθύμησαν ότι δεν είναι ικανοποιημένε με την κατανομή των ποσοστώσεων και ότι θέλουν να διαπραγματευτούν για να πετύχουν μεγαλύτερη ποσότητα. Ωστόσο, δεν παρουσίασαν επιχειρήματα δεν ε, παρουσίασαν καμία συγκεκριμένη ε, τοποθέτηση. Το μόνο που είπαν είναι ότι θέλουμε περισσότερη ποσόστοση και όχι το 5,16%. Συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Τον Ιανουάριο του 2013 ε, δεν προσχώρησαν οι νήσοι Φερόε στην συμφωνία για την κατανομή των ποσοστώσεων. Ήταν ξεκάθαρη η βούλησή τους. Ε, θα ξεκινούσε η αλευτική περίοδος και το μόνο, ο μόνος τρόπος που μπορούσαμε να προχωρήσουμε ήταν να έχουμε συμφωνία μεταξύ τεσσάρων μερών και να μείνουν οι νήσοι Φερόε έξω από την συμφωνία. Στη συμφωνία των τεσσάρων ε, η ποσόστοση των νήσων Φερόε παρέμεινε εκτός για το 2013. Τον Μάρτιο του 2013 ανακοίνωσαν οι νήσοι Φερόε την μονοπλευρή τους και μονομερή απόφαση να υιοθετήσουν ποσόστοση ύψους ε, που ανέρχεται στο 17% των μέγιστων επιτροπόμενων αλλιευμάτων έτσι όπως τα είχαν προτείνει οι ειδικοί για το 2013. Δηλαδή τριπλασίασαν, θέλησαν να τριπλασιάσουν την ποσόστοσή τους. Λοιπόν, η κατάσταση των αποθεμάτων Ρέγκας είναι πολύ ευάλωτη. Ξεκίνησαν να αυθύνουν τα αποθέματα ήδη από πέρσι και η τετραμερής συμφωνία μεταξύ των άλλων παράκτιων χωρών ε, περιλάμβανε μεγάλη δραστική μείωση της τάξης του 30% στη δυνατότητα αλίευσης των τεσσάρων αυτών μερών. Δηλαδή, όλα τα μέρη που είναι υπεύθυνα μειώνουν τις ε, ποσοστώσεις τους ο καθένας και ένα πέμπτο μέρος τριπλασιάζει τη δική του ποσόστοση. Αυτό δεν είναι ούτε υπεύθυνο ούτε λογικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε επανειλημμένως να πείσει τις νήσους Φερόε ότι δεν είναι σωστή αυτή η στάση αυτή την περίοδο και γι' αυτό ε, ήρθε σε επαφή με τη διοίκηση σε διάφορα επίπεδα, αλλά και με την πολιτική ηγεσία των νήσων, χωρίς όμως επιτυχία. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι θα έπρεπε να αξιοποιήσει τις ε, δυνατότητες ε, του κανονισμού 1026 του 2012, δηλαδή του κανονισμού που ασχολείται με τα επορικά εργαλεία. Περνάω λοιπόν τώρα στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου, να σας περιγράψω αυτά τα μέσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπεται λοιπόν στον κανονισμό 1026 του 2012, κοινοποίησε στις νήσους Φερόε ε, την πρόθεσή της να αναγνωρίσει τις νήσους αυτές ως ε, χώρα που, ε, στην οποία θα επιβληθούν αυτά τα εμπορικά μέτρα έδωσε στη χώρα αυτή η προθεσμία ενός μήνα για να απαντήσει. Στην ε, κοινοποίηση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε όλα τα επιχειρήματα που τεκμηριώνουν αυτή την απόφαση αυτής της την απόφαση αυτή της Επιτροπής ότι η Νίση Φερόε δηλαδή είναι μια χώρα η οποία αλλιεύει με μη υπεύθυνο τρόπο η Νίση Φερόε δεν απάντησαν με ικανοποιητικό τρόπο δεν απάντησαν ικανοποιητικά και η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία για τη λήψη αυτών των μέτρων τα οποία τελικά υιοθετήθηκαν στις 29 Αυγούστου δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα στις 21 Αυγούστου και άρχισαν να ισχύουν στις 28 Αυγούστου. Και Περί τίνος πρόκειται. Απαγόρευση ε, να μπει στην κοινοτική αγορά ρέγκα που έχει αλλιευθεί από τις νήσους Φερόε. Αλλά ε, και άλλα ψάρια που έχουν αλλιευθεί υπό τις ίδιες συνθήκες με την προσθήκη των άλλων ψαριών και πιο συγκεκριμένα ε, του σκουμπριού ε, πρέπει να σας πω ότι το σκουμπρί είναι, ε, αλλιεύεται παρεπιπτόντος όταν αλλιεύεται η ρέγκα. Και έτσι μέσω του σκουμπριού θα μπορούσαν ε, οι νήσοι Φερόε να εκμεταλλευτούν αυτό για να προωθήσουν επίσης ρέγκα. και γι' αυτό είναι παραλίευμα δηλαδή το σκουμπρί στη ρέγκα και γι' αυτό απαγορεύσαμε τις εισαγωγές στην κοινότητα αυτών των δύο ψαριών που έχουν ψαρέψει επιχειρήσεις αλλιευτικά σκάφη που ανήκουν στις νήσους και επίσης απαγορεύσαμε εκφόρτωση από αλληλευτικό στόλο των ίσων αυτών στα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πάλι για αυτά τα δύο ήχθη αποθέματα. Ε, ισχύει λοιπόν ο κανονισμός, εφαρμόζεται αυστηρά από τα κράτη-μέλη. Έχουμε ήδη ε, εξελίξεις και πληροφορίες ότι λειτουργεί ο κανονισμός αυτός Πάρα πολλά αλλιευτικά σκάφη ανησυχούν ιδιαιτέρως διότι δεν μεταφέρουν μόνο ρέγγα και σκουμπρί αλλά μεταφέρουν και άλλα εμπορεύματα. Είναι ε, φορτηγά πλοία, έχουν τεράστιες, ε, τεράστια χωρητικότητα, μεταφέρουν διάφορα άλλα εμπορεύματα και φρούτα, προκυπευτικά, άλλες προμήθειες δηλαδή. Επομένως, το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι αν μεταφέρουν ρέγγα ή σκουμπρί δεν θα μπορέσουν να μπουν σε κοινοτικό λιμένα και δεν θα τους επιτρεπεί να καταπλέψουν στο λιμένα, σίγουρα είναι κάτι που τους ε, κάνει να το σκέφτονται ε, δύο φορές, εάν θα δεχτούν να μεταφέρουν δηλαδή ρέγγα και σκουμπρί, γιατί πλήττονται και στα άλλα εμπορεύματα που μεταφέρουν. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό θα εξαναγκάσει τις νήσους Φερόε να υιοθετήσουν μια πιο ε, συμφιλιωτική ή συμβιβαστική στάση. Περνάω τώρα στο τρίτο μέρος της παρουσίασής μου και θα σας ε, παρουσιάσω την ε, τωρινή κατάσταση, το πώς έχει τα πράγματα με τις διαβουλεύσεις. Στόχος μας είναι αυτή η διαμάχη που έχουμε να αντιμετωπιστεί. Αλλά εμείς ποτέ δεν αρνηθήκαμε την συζήτηση, την διαβούλευση, όλα τα μέσα που θα βοηθούσαν να καταλήξουμε σε συμφωνία. Η Κομισιόν λοιπόν μαζί με τις νήσους συναντήθηκαν εκ νέου στο Λονδίνο 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Στη συνεδρίαση αυτή δυστυχώς για άλλη μια φορά τα νησιά Φερόε δεν έδειξαν ε, καλή θέληση, σαφή θέληση να διαπραγματευτούν. Παρ' όλα αυτά σημειώθηκαν μικρές προόδοι, συμφωνήθηκε δηλαδή να δημιουργηθεί μια επιστημονική ομάδα εργασίας που στο μέλλον θα επέτρεπε να εντοπίζονται καλύτερα τα βιογεωγραφικά δεδομένα που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν καλύτερα στην κατανομή των αλλιευμάτων στο μέλλον. Στη συνάντηση αυτή όλοι οι άλλοι εκτός από τις Φαρόες συμφώνησαν ότι για το 2014 πρέπει να συνεχιστεί η κλίδα κατανομής που αποφασίστηκε το 2007 μέχρι να καταλήξουμε σε νέα συμφωνία. Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα ότι οι νήσοι Φερόε με τη στάση τους δεν δείχνουν να έχουν σαφή βούληση να υπάρξει συμφωνία αλλά προσπαθούν να κολυσιεργήσουν όσο γίνεται την εξέβρεση λύσης. Τέλος. Α, όχι. Α, α συγγνώμη. Επίσης, τονίζω ότι Σήμερα, σήμερα, τα 11 παράκτια κράτη συνεχίζουν να συζητούν τις δυνατότητες αλληλείας για το 2014. Δεν έχω πληροφόρηση γιατί τώρα γίνεται η συνάντηση για το εάν θα υπάρξει συμφωνία το 2014. Η Κομισιόν είναι δεδεθειμένη να διαπραγματευτεί, είναι δεδεθειμένη να κάνει και παραχωρήσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Αυτά τα, αυτές τις εμπορικές κυρώσεις ε, ε, τις κάναμε μόνο και μόνο ως εισαγωγική κίνηση. Τώρα για την διαδικασία διατησίας. Στις 21 Αυγούστου, που ήταν η μέρα που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα, ή εμπορικές κυρώσεις. Ε, στη, στη Δανία υποβλήθηκε έτοιμα από τις Φερόες να αρχίσει η διαδικασία διαιτησίας με βάση τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σε αυτήν την ενημέρωση οι Φερόες ζήτησαν να δημιουργηθεί ένα ε, ε σώμα διατησίας που να αντιμετωπίσει τη καταγγελία από τις Φερόες των Φερόων ότι έχει, ότι έχει παραβιαστεί το άρθρο 63 παράγραφος 1 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσης και ζητούσαν η Επιτροπή να σταματήσει την επιβολή κατασταλτικών όπως αποκαλούν μέτρων διότι κατά τη γνώμη των Φαροών αποτελούν διακρίσεις που στόχο έχουν να επιβάλλουν κατανομή υπέρ της Ένωσης, προς το συμφέρον της Ένωσης και άρα δυσχεραίνουν την εξέβρεση λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων. Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η διαδικασία διατησίας που προτείνουν οι Φερόες δεν ε, επιχειρεί καν να λύσει το θέμα της ουσίας την κατανομή των αποθεμάτων Ρέγκας. Αυτό που επιδιώκει αποκλειστικά αυτό το αίτημα είναι να σταματήσουν τα εμπορικά μέτρα, διότι θεωρούν ότι έτσι παραβιάζεται ε, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, γιατί θεωρούν ότι είναι κατασταλτικά αυτά τα μέτρα. Η Επιτροπή απάντησε σε αυτήν την ανακοίνωση των ε, Φερών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Να σε εξηγήσω τώρα λίγο πώς είναι η διαδικασία. Πώς λειτουργεί από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ειδοποίηση. Στην ειδοποίηση των φαρών προτείνεται ποιο μέλος του σώματος διατησίας πρέπει να διοριστεί λέγεται ότι με βάση την διαδικασία ότι για αυτό το σώμα ε, ε, επιδιαιτησίας ο καθένας ο καθένας, το κάθε εμπλεκόμενο μέρος προτείνει έναν ε, εκπρόσωπο, ένα διαιτητή. Πρότειναν τον κύριο Ουκούνια, ο οποίος είναι από τη Χιλή, πολύ διακεκριμένος νομικός. Η Κομισιόν επίσης πρότειναν πολύ διακεκριμένο ε, Νομομαθεί από την Αυστρία, τον κύριο Ζεράρ Γκέρχαρτ Χάφνερ. Η επόμενη φάση της διαδικασίας είναι ότι άλλα τρία μέλη αυτού του σώματος πρέπει να ε, διοριστούν συνενετικά. Η Κομισιόν ε, ρώτησε το Συμβούλιο, το Συμβούλιο πρότεινε μια σειρά από ονόματα και έγινε η πρώτη συνάντηση με τις Φερόες που δεν κατέληξε συνεχίζονται διαβουλεύσεις για να μπορέσει να συσταθεί σε σώμα αυτό το σώμα επιδιαιτησίας. Συνήθως προβλέπονται από τη στιγμή της ε, ειδοποίησης 60 μέρες για να συσταθεί αυτό το σώμα, άρα θα έπρεπε στις 21 Οκτωβρίου. Εάν δεν συμφωνούν βέβαια οι εμπλεκόμενοι, για την ε, σύνθεση του σώματος, τότε το ε, δικαστήριο για το δίκαιο της θάλασσας, ο πρόεδρός του συγκεκριμένα, αποφασίζει τα τρία, για τα τρία μέλη, τα τρία υπόλοιπα μέλη του σώματος επιδιαιτησίας αυτού. Πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν στην απάντησή της στην ειδοποίηση της Δανίας δέχτηκε αυτή τη διαδικασία επιδιαιτησίας διότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Όταν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε το δίκαιο της θάλασσας, δεν ε, πρότεινε συγκεκριμένη διαδικασία για την επίλυση διαμαχών, οπότε ελήψη άλλης ε, διάταξης είναι αυτό που προβλέπει η σύμβαση. Η διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική. Δηλαδή, αν ένα τμήμα κάνει επίκληση αυτής της διαδικασίας διατησίας, προχωράει η διαδικασία ανεξάρτητα από το εάν συμφωνεί το άλλο εμπλεκόμενο τμήμα. Ακόμη και αν η Κομισιόν λοιπόν δεν αποδεχθεί τη διατησία, εφόσον είναι η μόνη διαδικασία που προβλέπεται, θα συνεχίσει την πορεία της αυτή διαδικασία. Και θα συνεχιζόταν αυτή η διαδικασία χωρίς να ακουστεί στα πλαίσια της διαδικασίας η άποψη της Ένωσης. Άρα ε, πρέπει να δεχθούμε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να σας πω ότι η διαδικασία αυτή και ακόμη περισσότερο η απόφαση της διατησίας είναι υποχρεωτική. Για τις άλλες περιπτώσεις, ξέρετε, ε, η διαδικασία διατησίας κάνει συστάσεις. Εάν υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία απόφαση της διατησίας, είναι δεσμευτική. Να μην πω άλλα. Απλώς να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή ακόμη λοιπόν προσπαθούμε να καθορίσουμε τη σύνθεσή του και στη συνέχεια αυτό το σώμα επιδιαιτησίας θα καθορίσει τη διαδικασία του, ε, το χρονοδιάγραμμα εργασιών του. Το πώς θα εκτελέσει το καθήκον του. Το κόστος ε, το φέρουν ε, οι διάδικοι. Η Κομισιόν εκπροσωπεί την Ένωση αυτή τη διαδικασία. Ελπίζουμε να ενημερώσουμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για το πώς προχωράει η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Λοιπόν, πρώτος ο κύριος Γκάλαχερ. Κατά πρώτον, Πρόεδρε, να πω ότι το ενημερωτικό σημείο που μιλάβαμε ήταν πολύ λεπτομερές και διαφωτιστικό. Νόμιζα όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το σκουμπρί και την Ισλανδία θα έκανε κάτι συγκεκριμένο. Την ξέραμε την όλη διαδικασία την πρώτη φορά που χρειάστηκε να εφαρμοστεί. Τότε που έλαβε τα απαραίτητα βήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέσα 2050 και την έκθεση που είχε εγκρίνει το Κοινοβούλιο σχεδόν ομόφωνα. Νομίζω έξι μέλη του Κοινοβουλίου καταψήφισαν τότε και αυτό ήταν σχεδόν αποσφάλμα. Ε, θα λέγαμε το 100% υπερψήφισε. Πέραν όλων αυτών, αυτό που κατανοώ είναι ότι αυτή η διαιτησία δεν ασχολείται με την ουσία του προβλήματος. Απλώς κοιτάζει τι βήματα έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι κατά πόσον έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ότι δηλαδή δεν θα έπρεπε να εισάγεται το σκουμπρί ή η, η ρέγγα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως θέλει να ελέγξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα δεν ήταν αυστηρά, αλλά έτσι κι αλλιώς ελπίζουμε ότι αφού δήλωσε η Επίτροπος ε, ξεκάθαρα στην Επιτροπή Αλίας και προς το τέλος του Ιουλίου πριν την διακοπή για το καλοκαίρι ότι τα ίδια μέτρα θα προβλέπονταν κατά της Ισλανδίας και των Φερών για την υπεραλίευση του, του σκουμπιού. Εδώ πρέπει να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εκτιμήσαμε πολύ την παρουσία της ίδιας της Επιτρόπου εδώ και όσα μας είπε. Αλλά ίσως ήταν απλουστευτική αυτή η άποψη. Είναι πολύ έξυπνη η κίνηση το Ισλανδίας των διότι Συναντηθήκαμε στο Λονδίνο πρόσφατα και ζήτησαν από επιστημονικό σώμα και περισσότερα στοιχεία και πιέζουν, πιέζουν ε, με επιτυχία. Εάν είχαμε άλλο κοινοβούλιο ή άλλη επίτροπο θα είχαμε χάσει να, στην προσπάθεια να ελέγξουμε την αλίευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε από το παρελθόν μια ε, διακρατική συμφωνία και θα έπρεπε να ισχύσει. Αλλά αυτά έχει η διατησία. Και τι είναι αυτή η διατησία. Μιλάμε για 5,6% αλίευση το 2012 και έχουμε φτάσει στο 17% τώρα. Μα δεν θέλαμε αυτό. Αυτό που θέλαμε είναι μέτρα που νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση τα είχε λάβει. Τα είχε λάβει εντός των κριτηρίων που προέβλεπε ο νόμος. Ε, όμως ήθελα να καταλάβω τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει συμβούλιο στο Λουξεμβούργο και με απασχολεί αν η Επιτροπή σκέφτεται να κάνει παραχωρήσεις στις Φερόες και στα 11-12% για το σκουμπρί και στην Ισλανδία 11,9. Ε, Πέραν αυτού, η Ρωσία και η Γρυλανδία θα προσθεθούν σε αυτή τη συμφωνία. Πολλές παραχωρήσεις. Η ISIS πρότεινε αύξηση 64% για την ποσόστοση του σκουμπρίου φέτος στο Βορειοατλαντικό. Γιατί, γιατί τα ευρωπαϊκά σκάφη έδειξαν ε, ανεύθυνη στάση. Πέρσι όμως ήταν 150.000 η συνολική ποσόστοση για τα κράτη του Βόρειου Ατλαντικού. Και όποια και αν ήταν η φόρμουλα που τελικά θα επιλέγαμε, δεν πρόκειται να το πετύχουμε. 150. Από αυτή την ε, δεξαμενή δυνατοτήτων βγάλαμε 150, ε, ένα εκατομμύριο τόνους. 150.000 τόνοι λοιπόν πρόσθετο από το σύνολο που είχαμε. Τα ίδια όπως πριν από δεκαετία που είχαμε πρόβλημα με το προσφυγάκι. Και πέραν αυτών, ναι, πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς στιγμή προσπαθεί να ε, κάνει συμφωνίες με τις υπόλοιπες χώρες για να τις πάρει με το μέρος της χώρες που εξαρτώνται από τα σκουμπρί και τα άλλα είδη, τα πελαγικά. Αυτές οι χώρες τηρούν υπεύθυνη στάση. Και είδαμε τους τελευταίους μήνες ότι 35% των αποθεμάτων που έλεγαν Ισλανδοί ότι βρίσκονται στα ύδατα της Ισλανδίας έχουν περάσει στα ευρωπαϊκά. Δεν πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε ούτε να, συγκατα... να είμαστε συγκαταβατικοί σε οποιαδήποτε παραχώρηση μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να επιμείνουμε και να είμαστε σκληροί στη στάση μας στις διαπραγματεύσεις. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα η παρέμβαση του κ. Κόβνη, του πρώην Πρόεδρου του Συμβουλίου, θα μπορέσει να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Εγώ έθεσα το ερώτημα και δεν ήθελα να είμαι προκλητικός, αλλά πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επίτροπο, εκπροσωπούν τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προασπίζονται με τον καλύτερο τρόπο, ή τελικά του επιτρέπουμε να ελίσσονται και μέσα από αυτό τον. Ε, μέσα από τους διάφορους ελιγμούς τους να κερδίζουν χρόνο και τους επόμενους μήνες. Έχω και μια σειρά από άλλες παρατηρήσεις, αλλά τι γίνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τι συμβαίνει. τα λάθη και τις κακές κινήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες. Τέλος πάντων, εγώ ανησυχώ ιδιαιτέρως. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μένω ο θεματοφυλακάς μας, αλλά στο τέλος θα στραφούμε στη Νορβηγία για να σώσει τα πελαγικά είδη και την αλία, την αλία τους ε, για τα ευρωπαϊκά σκάφη. Πραγματικά ε, θα το πω ε, στην ε, Επίτροπο και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να τη το εκφράσει. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από το Κοινοβούλιο με τη στάση τη. Μα τα είπε τον Ιούλιο και τώρα ξεκινάει η διαδικασία που είναι γνωστή ω κινητοποίηση του εμπορικού εργαλείου. Τίποτα δεν έχει γίνει από τον Ιούλιο. Δεν μπορούμε να βρούμε καν την Επίτροπο. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον από την Επιτροπή να έρθει να μα μιλήσει. Κάτι πρέπει να καταφέρουμε εδώ Βλέπω ότι το σημείο 11 μιλά για δράσεις που έχουν αναλυφθεί κατά της Ισλανδίας και των Φερών. Εδώ δεν έχει γίνει τίποτα. Μόνο για τη Σκανδιναβία έχουν ληφθεί μέτρα. Με τη Σκάνδια και την Άβο. Ε... Ευχαριστούμε κυρία Λέβιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Η ερώτησή σας, Πρόεδρε, είναι πολύ εύστοχη. Uh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική της παρουσίαση και τις δηλώσεις της. Νομίζω ήταν, ε, συναρπαστικό, ήταν συναρπαστικά όσα ακούσαμε και ήταν ε, ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Μιλάμε για κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε πολλές περιοχές του κόσμου, ούτως ή άλλως στο μέλλον. Δεν είναι η το, το τι γίνεται με τα μεταναστευτικά ήδη αυτό που μας απασχολεί, αλλά και κλιματικές αλλαγές και εξελίξεις που προκύπτουν από αυτές. Ε, μιλάμε για κοινά αποθέματα σε πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι λοιπόν τόσο σαφές ε, να μπορεί να πει κανείς ότι είναι όλα μαύρα ή άσπρα, πρόκειται για ευρωπαϊκό απόθεμα ή ισλανδικό. Ε, πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας αυτά, θα τα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Έχω όμως λίγες ερωτήσεις. Πρώτον, εάν σωστά κατάλαβα, η, τετραπλή συμφωνία η οποία συνεχίστηκε στην αρχή της χρονιάς δεν συμπεριλαμβάνει τις Φερόες. Ε, τους έχει αποδοθεί ποσό στο ΣΥΤΑΚ ή όχι. Μετά, σε ό,τι αφορά τα δεδομένα για τις ε, επιπτώσεις στην οικονομία των ε, νήσων, λόγω της ε, θέσης σε ισχύ της απαγόρευσης εισαγωγής ρέγκας και παρόμοιων ειδών. Άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρόλο που υπάρχουν ε, και άλλα είδη φορτίου, ε, τελικά αυτά δεν μπορούν να περάσουν λόγω της παρουσίας ρέγκας στα ευρωπαϊκά ύδατα. Φαντάζομαι ότι έχουν πληγεί άσχημα οι φερόες από αυτόν τον κανονισμό. Επίσης, το 40-50% είναι τεράστιος αριθμό για το εξαγωγικό εισόδημα των φερών. Ε, ε, στα ψάρια βασίζονται. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σοβαρό ο αντίκτυπος ε, για αυτούς. Τι γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το βαθμό στον οποίο έχουν πληγεί ως τώρα. Μετά το θέμα για τι φερόε που θα προσάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο διαιτητικό όργανο του ΟΗΕ. Θα κινητοποιηθούν, από ό,τι φαίνεται, οι μηχανισμοί διατησίας του άρχους. Αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και δεν ξέρω πόσες φορές έχει γίνει κάτι τέτοιο στο παρελθόν, αλλά ξέρω ότι οι Φερόες είναι σε πολύ ε, δυσμενή θέση ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζήτησε από μόνη της ε, διατησία. Και ανταυτού έλαβε μέτρα τα οποία τα θεωρούν ιδιαίτερα εχθρικά. Η ερώτηση λοιπόν είναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτηκε σε κάποια περίπτωση να το δει αυτό μαζί με τα άλλα παράκτια κράτη, διότι δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα. Τολμώ να πω ότι πρόκειται για ένα κοινό. Μάλλον είναι ε, μια κοινή αντίληψη για τις ε, Φεροές ότι η ποσόστοση ε, επιβλήθη μονομερώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Η Ισλανδία και η Νορβηγία συμμετείχαν στην επιβολή της ποσόστοσης. Και αυτό ε, για να απαντήσουν στην, στον τριπλασιασμό, το μονομερή τριπλασιασμό από την πλευρά των φερών. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, έλαβε, ποτέ, σκέφτηκε ποτέ μεταξύ των άλλων επιλογών να κάνει κάτι. Θα ήθελα να το ακούσω και αυτό και να μου πείτε την άποψή σας. Συμφωνώ απολύτως ότι οι θερόες. Είναι κάπως άκαμπτη στις διαδικασίες, στις διαπραγματεύσεις, όμως νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Η κατανομή της ρέγκας και του σκουμπριού όντως μπορεί να έχει αλλάξει. Πρέπει να βασίσουμε την αποτίμησή μας στην επιστημονική αλήθεια, στα επιστημονικά πορίσματα. Η κλίδα κατανομής που χρησιμοποιούμε σήμερα μπορεί να μην είναι σκοπιμότερη. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε εάν χρειάζεται μια νέα κλίδα κατανομής που να απηχεί και την πραγματική παρουσία των ψαριών. Πώς κατανέμονται αναγεωγραφικά και συντεταγμένε και ούτω καθεξή. Η άποψή μου είναι ότι τα ηχθικά από θέματα, εφόσον είναι κοινά, πρέπει να είναι και αντικείμενο βιώσιμη διαχείριση. Από κοινού. Ότι όλα τα μέρη πρέπει να αναλαμβάνουν τι ευθύνε του. Η Ισλανδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Φερόε, η Νορβηγία, όλοι μαζί. Δεν ανήκουν σε κανέναν αποκλειστικά. Δεν τα βάλαμε εμεί στο νερό τα ψάρια. Εκεί ήταν από πριν. Είναι πραγματική πόρη. Επίσης θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι που φαίνεται να έχει ξαφνιάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, τους, και όλους. Τι είναι αυτό το διαιτητικό δικαστήριο. Πού υποτίθεται ότι θα τα συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά. Και αυτό πώς θα επηρεάσει το νέο μας κανονισμό. Περί απαγόρευσης εισαγωγών από χώρε που επιτρέπουν την ίδια όσημη αλίευση δεν είναι σαν να λέμε, μάλλον ο σωστός τρόπος δεν θα ήταν να περάσουμε από το διαιτητικό όργανο του ΟΗΕ και να δεχτούμε τη δική τους απόφαση. Γιατί να επιβάλλουμε μπορικές κυρώσεις. Όπως είπε και ο Άγγους, πρέπει να σκεφτούμε κάθε δυνατή επιλογή για να φτάσουμε σε συμφωνία, προτού έχουμε και σοβαρότερες κυρώσεις και αντίπεινα μεταξύ μας. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπω και ο Πάτρικ. Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο εδώ, ε, αν είναι δίκιο αυτό που κάνουν οι Φερόες ή εμείς αυτούς. Και για την Ισλαμπία το ίδιο. Αλλά θα ήθελα να συγκεντρωθώ στις Φερόες τώρα. Ε, για μένα δεν είναι σαφές από όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το άκουσα, ότι οι Φερόες επανειλημμένως δεν έχουν αιτιολογήσει, δεν έχουν εξηγήσει γιατί απαιτούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα αλλιεύματα. Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο. Αν είχαμε εδώ κανέναν εκπρόσωπο των φερών. δεν μπορεί να μας λένε απλώς θέλουμε κι άλλα. Θέλουμε κι άλλα γιατί υπάρχουν πιο πολλά ψάρια, εντάξει. Ή δεν τα είχατε κατανείμει δικαίως του παρελθόν, εντάξει. Αλλά κάτι, να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Να καταλάβουμε γιατί τα λένε αυτά που λένε. Θα ήθελα κάποιο σχόλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταλάβω που προέκυψε όλη αυτή η στάση. Αλλιώ θα πρέπει να κοιτάξουμε πώ έχει η κατάσταση των αποθεμάτων σήμερα και πώ ε, έχουν αλλάξει από το 2007 και πώ έχουν καταναμηθεί από το 2007 σήμερα. Και μετά, ποιε είναι οι πολιτικέ συνέπειε όλων αυτών ακούσαμε ότι οι εξαγωγές ε, ψαριών ρέγκας και σκουμπιού είναι τεράστια σημασία για την οικονομία των θερών. Είναι κινητήριος δύναμη της οικονομίας τους. Αλλά τι εννοούμε εδώ, ότι υπάρχουν αργοκίνητα σκάφη που ε, κυνηγάνε μόνα τους τις ρέγγες και τις ψαρεύουν ή είναι τίποτα μεγάλες εταιρείε, μια-δυο μεγάλες εταιρείε που πιέζουν, πιέζουν για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Και ε, μέσα σε αυτή την πολιτική στάση την Φερών, τι ε, απόϊχος υπάρχει από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας εκεί ή από τους πολιτικούς τους. Τι δυνατότητα μπορεί να υπάρχει για τις διαπραγματεύσεις να α, ε, μεταβάλλουν τη στάση τους. Και για τη διαδικασία διατησίας ποιος ε, την πληρώνει. Είναι τρομεροί οι δικηγόροι που έρχονται, αλλά μπορεί να κοστίσουν περισσότερο από την παραχώρηση της ποσοστοσή για τη ρέντα. Θέλουμε απλώς να κατανοήσουμε καλύτερα και την άλλη πλευρά. Αυτό είναι όλο. Κυρία Λέβιν, ευχαριστώ. Ενημερωθήκαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ε, επιπλέον αλίας στις Φερόες έχει αναλάβει Ολλανδική εταιρεία. Το χρήμα ρέει και πάλι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ίσως να ξέρει περισσότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Ευχαριστούμε και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω καταρχάς στην ερώτηση του κυρίου Γκάλαχερ. Τι γίνεται με το σκουμπρί και τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το σκουμπρί και την Ισλανδία. Θα θυμάστε ότι τον Απρίλιο έγιναν εκλογές στην Ισλανδία, σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση τον Μάιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή πριν αναλάβει, οποιαδήποτε δράση να δώσει μια ευκαιρία στη νέα κυβέρνηση να αλλάξει στάση ως προς το σκουμπρί. Η Επίτροπος κυρία Δαμανάκη είδε τον Υπουργό Αλληλείας στις αρχές Ιουνίου και δεν ε, είδε να αλλάζει η στάση της Ισλανδίας καθόλου. Ωστόσο, κατέστησε σαφές στις, ε, στους νέους πολιτικούς ηθήνοντες της Ισλανδίας ε, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Επίτροπος είπε ξεκάθαρα ότι θα εκτελέσει την εντολή των κρατών μελών και το αίτημα άλλωστε μέλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αξιοποιηθούν οι εμπορικές κυρώσεις ως εργαλείο, ως μέσο εκτός και αν αλλάξει η στάση της Ισλανδίας. Τα κατέστησε όλα αυτά σαφή και έκτοτε υπήρξαν κάποιες επαφές με την Ισλανδία, όχι πολύ πιστικές, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την διαμόρφωση της ε, επιχειρηματολογίας η οποία θα συνταχθεί στην γνωστοποίηση που θα αποσταλεί στην Ισλανδία. Ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πρόθεση να χαρακτηρίσει την Ισλανδία ως χώρα που ε, κάνει μία υφόρο αλληλευτική δραστηριότητα και άρα θα υπόκειται στις εμπορικές κυρώσεις ή μέτρα. Και όλα αυτά συνέπεσαν με μία αλλαγή πολύ σημαντική της κατάστασης. Ποια είναι αυτή? Ο, ολοκληρώθηκαν οι εκστρατείες των σκανδιναβικών χωρών με τις ε, ε, νήσους Φερόε και την Ισλανδία και με την ε, συμβολή Ευρωπαίων επιστημόνων Όλη αυτή η επιστημονική εκστρατεία κατέληξε στο πόρισμα ότι το απόθεμα σκουμπριού αυξάνεται και μάλιστα με θεαματικό τρόπο. Η τελευταία συνεδρίαση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εκμετάλλευση της Θάλασσας έλαβε χώρα τον Αύγουστο και επιβεβαίωσε του λόγου το αληθές. Επιβεβαίωσε την ε, ε, επιστημονική άποψη λοιπόν. και φαίνεται ότι πράγματι είχε αυξηθεί το απόθεμα σκουμπριού και μάλιστα με θεαματικό τρόπο. Με, ε, φάνηκε αυτό και από την επιστημονική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οτοκία. Θεωρούμε μέχρι αυτή τη στιγμή ότι η υπεραλίευση Ισλανδίας και νήσων Φερόε έκαναν τα ηχθιαποθέματα να μειωθούν και μάλιστα να πέσουν κάτω από το επίπεδο της ε, ε, μέγιστης αηφόρου απόδοσης. Και ότι δεν πληρείται το κριτήριο για να θεωρηθεί η χώρα αυτή ως ασκούσα μια αλληλευτική δραστηριότητα ε, μη βιώσιμη σε σχέση πάντοτε με το 2013. Άρα κατέπεσε το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, χρειαζόταν η Επιτροπή νέα επιχείρηματα για να ε, προσφύγει εναντίον των χωρών αυτών στη χρήση αυτών των μέσων και κυρώσεων. Αυτό από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, το ότι άλλαξε η κατάσταση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία. Γιατί το λέω αυτό. Διότι ε, εάν οι τεράστιες θυσίες, η μείωση των ελευτικών δυνατοτήτων ε, μπορεί να έχουν γίνει, δηλαδή δεν ζητάτε μείωση ελευτικής ε, δυνατότητας. Είναι ευκαιρία λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερη κατανομή, γιατί όταν η πίτα είναι μεγαλύτερη, είναι μεγαλύτερο και το κομμάτι που θα πάρει ο καθένας. Και γι' αυτό η Επιτροπή έδωσε προτεραιότητα στο εξή. Αξιοποίησε όλες τις δυνατότητες για να πετύχει συμφωνία πριν το 2014 και έδωσε προτεραιότητα σε αυτή τη διαδικασία και όχι τόσο στην υιοθέτηση των εμπορικών ε, κυρώσεων ή μέτρων. Διότι θα ήταν μάλλον απίθανο να το πετύχει, γιατί δεν ε, πληρεί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως μη βιώσιμα αλληλεία, η αλληλεία αυτών των χωρών. Η κυρία Λέβιν λοιπόν έκανε πολλές συγκεκριμένες προτάσεις. Πρώτο, για την τετραμερή συμφωνία και αν περιλάμβανε τις νήσους Φερόε, απαντώ και λέω όχι. Η συμφωνία των τεσσάρων μερών επετεύθη, εγκρίθηκε, να μην πω κυρώθηκε, ούτε καν συμφωνία. Αλλά, εν αυτές οι διαβουλεύσεις κατέληξαν σε αυτή τη διευθέτηση, η οποία εγκρίθηκε και συμφωνήθηκε είναι ένα arrangement, μια διευθέτηση. Δεν είναι δεσμευτική νομικός συμφωνία, είναι μια συμφωνία κυρίων επί της αρχής η οποία δεσμεύει τα μέρη που κάθονται γύρω από το τραπέζι. Δηλαδή, αυτά θα συστήσουν στους ηθήνοντές τους και στους ανωτέρους τους την αντίστοιχη λήψη μέτρων. Αυτή η ανεπίσημη λοιπόν διευθέτηση συμφωνία δεν περιλάμβανε τις νήσους Φερόε γιατί δεν θέλησαν να μπουν σε αυτήν. Αλλά αυτό το οποίο πράγματι εγκρίθηκε και συμφωνήθηκε ήταν το εξή. Από το μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα για το 2013 να αφήσουμε κατά μέρο την ποσόστοση που θα αντιστοιχούσε στις νήσους Φερόε και να κατανείμουμε μόνο το υπόλοιπο μεταξύ των τεσσάρων μερών. Η κυρία Λέβιν επίσης ρώτησε το εξής. Αν έχουμε στοιχεία για οικονομικά για τις νήσους Φερόες. Δεν τα έχουμε. Ίσως ε, τα ίδια τα νησιά από μόνα τους κάνουν μια τέτοια αξιολογήση. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ε, επικοινωνιακή τους εκστρατεία. Εμάς δεν μας αφορά. Ή μπορούν να το μεγιστοποιήσουν και να πούνε βεβαίως και μας αναφορά υπέστημαν ε, μεγάλο πλήγμα από την ε, καταπίεση του Γολιάθ που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία επιτίθεται στον ε, μικρό Δαβίδ. Δεν ξέρουμε επικοινωνιακά πώς θα το χειριστούν. Και απαντώ και στο τρίτο σας ερώτημα ή μάλλον στο ερώτημα του κυρίου Ντέιβις εάν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδρασή τους. Στον τύπο έγινε, δεν έγινε μεγάλος λόγος για αυτό το θέμα. Ελάχιστα είναι τα δημοσιεύματα και δεν είναι βέβαια πολύ ικανοποιημένοι, αυτό το γνωρίζουμε. Η άποψη του πληθυσμού ήταν εξαιρετικά αρνητική και η κυβέρνηση ανησυχεί ιδιαίτερως με τον αντίκτυπο αυτών των εμπορικών κυρώσεων και μέτρων. Η κυρία Λέβιν αναφέρθηκε στην ανάγκη εξάντλησης όλων των διαδικασιών ε, συμβιβασμού και συνδιαλλαγής μέχρι ότου υιοθετηθούν τα, οι εμπορικές κυρώσεις και πριν υιοθετηθούν αυτές. Συμφωνούμε. Απολύτως. Ωστόσο, ως προς τη Ρέγκα είναι πολύ επίγουσα η κατάσταση. Είναι πήγον το θέμα. Το απόθεμα εξαντλείται. Είναι πολύ κάτω από την μέγιστη αηφόρο απόδοση λόγω της υπεραλίευσης που έχει γίνει και θα υπάρξει υπεραλίευση και φέτος αναπόφευκτα. Θα πέσει ακόμα πιο χαμηλά ε, το απόθεμα αυτό και τα επιστημονικά πορίσματα το επιβεβαιώνουν αυτό, τα ηχθιαποθέματα κατα καταραίων και θα πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα. Ξέρετε, μια διαδικασία συνδιαλλαγής ε, μπορεί να κρατήσει από μήνες μέχρι και χρόνια. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Πρέπει να ληφθούν μέτρα αμέσως για να αντιμετωπιστεί η υπεραλήψη, να αποκατασταθεί το απόθεμα. Τα πέντε μέρη είχαν συμφωνήσει πάνω σε μηχανισμούς ανάκτησης αποθέματος και αν εφαρμοστούν αυτά πολύ γρήγορα θα, ανακάμψει, ε, θα ανακάμψουν τα ίχθη αποθέματα. Η κυρία Λέβιν τόνισε επίση το σημαντικό, ότι δηλαδή το σημαντικό είναι η αηφορία των αποθεμάτων. Συμφωνούμε απολύτω, προφανώς, και γι' αυτό ζητούμε άμεση και γρήγορη δράση. <coughs> Κύριε Ντέιβις, νέο καθεστώς για την κατανομή, τη διανομή της ρέγκα ή του σκουμπριού, αν υπάρχει ένα νέο ε, καθεστώς, το οποίο κάνει ε, αυτά τα είδη να εντοπίζονται περισσότερο στην Ισλανδία ή στις νήσους Φερόες. Ως προς το σκουμπρί αυτό έχει επιβεβαιωθεί, δηλαδή πολύ περισσότερα σκουμπρία υπάρχουν σε αυτή την περιοχή συγκριτικά με τα αποθέματα πριν το 2009, ε, οι νήσοι Φερόες και η Ισλανδία έχουν πολύ μεγαλύτερα αποθέματα σκουμπριού από ό,τι είχαν στο παρελθόν. Τεράστια διαφορά και αυτό είναι απτό, είναι, φαίνεται. Άρα πρέπει να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα αυτών των κρατών να αποκτήσουν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας αυτής. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα της Ισλανδίας, η οποία μέχρι πολύ πρόσφατα δεν ήταν μέρος των ε, παράκτιων κρατών. Θέλησε να αυτό χαρακτηριστεί ως παράκτια χώρα και να απολαύσει όλα τα δικαιώματα που συνεπάγεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Οι νήσοι έχουν δικαίωμα η κατανομή των αποθεμάτων να είναι ε, διαφορετική. Τώρα, ποιοι στόλοι ψαρεύουν. Τη Ρέγκα, στις νήσους Φερόες ψαρεύουν τη Ρέγκα τα ίδια σκάφη. Αυτά που ψαρεύουν Ρέγκα ψαρεύουν και σκουμπρί. Ίδιος είναι ο στόλος. Και δεν είναι μόνο στόλος ε, που φέρει σημαία των νήσων Φερόες είναι και στόλοι ελευτικοί που έχουν μισθωθεί, να βλωθεί από την κυβέρνηση ή από τις εταιρείες των νήσων Φερόε και φέρουν σημαία κινέζικη ενίοτε ή από το Περού και όταν αλλιεύουν στα ύδατα των ίσων φερόες δεν υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν αυτό στην ΑΝΕΑΣΚΕ και άρα δεν το μαθαίνουμε δια της άμεσης οδού. Η κυρία Λέβιν είπε ότι είχαμε και σκάφη με Ολλανδική σημαία. Είναι πιθανό αυτό, αλλά δεν το πιστεύω εγώ προσωπικά. Ορισμένα από αυτά τα σκάφη των ίσων Φερόες ε, τον ε, με κινέζικη σημαία ή με σημαία ε, Περού μπορεί στο μετοχικό τους κεφάλαιο να είναι κάτοχοι μέρους του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών που διαχειρίζονται αυτά τα σκάφη επιχειρήσεις ή άνθρωποι ευρωπαϊκής υπηκότητας αν θέλετε, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Τώρα, ποιος πληρώνει για όλα αυτά. Υπάρχει διαδικασία για τις δικαστικές διαμάχες. Πάντοτε υπάρχει κοινοτικός προϋπολογισμός, τμήμα του προϋπολογισμού που έχει τεθεί κατά μέρος για τέτοιου είδους διενέξεις και διαμάχες και θα αξιοποιηθούν αυτά τα κονδύλια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλαχερ. Καλά προωτήσαμε για το σκουμπρί, γιατί δεν ήταν τμήμα της αρχικής ερώτησης. Τη αρχικής παρουσίαση, αλλά δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Δεν θέλω να κατηγορήσω την Επιτροπή. Ε, μπορεί να ήταν τακτική τους, να τους πούμε ό,τι λιγότερο μπορούμε. Τώρα ξέρουμε την κατάσταση και οι χειρότεροι φόβοι μου επιβεβαιώνονται. Ποιοι είναι αυτοί. Λόγω του ότι η Ένωση έδρασε με υπεύθυνο τρόπο, τα μέτρα που πήρε η Ένωση, παραθέτω, βοήθησαν να ανακάψουν, να ανακάψουν τα λιεύματα, Ανέκαμψαν λοιπόν τα αποθέματα. Άρα, εφόσον υπάρχουν περισσότερα ψάρια, ας τα δώσουμε ε, και θα λύσουμε το πρόβλημα. Αυτή είναι η απάντηση. Χώρες που ε, πριν από χρόνια αλλιεύαν το 2,5% τώρα αλλιεύουν το 20%. Δηλαδή, όποιος δρά ανεύθυνα αμείβεται. Θα έπρεπε να εφαρμόσουμε τον απλό κανόνα ότι αν, αρχίζουν, αν ε, αυξάνονται τα τελικά αλλιεύματα, τα τωρινά αλλιεύματα, η κατανομή θα πρέπει να μείνει η ίδια. Γιατί να αυξήσουμε το ποσοστό πάνω από 600, να το αυξήσουμε για να αποφελθούν όλοι αλλά ελπίζω η απόφαση αυτή που δεν θα πάρουμε εμείς εδώ να μην ληφθεί και στο Λουξεμβούργο. Αλλά να πούμε ότι η Κομισιόν άλλαξε άποψη μετά τη δεύτερη ή τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου, τότε που είχαν πει ότι θα εφαρμόσουν τα εμπορικά μέτρα μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν περισσότερα αλλιεύματα. Είναι υπεύθυνη η αντιμετώπιση αυτή. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ξέρω ότι εσείς εδώ είστε πεισμένοι για αυτά που λέω, αλλά είναι κόλαφος για τα μέλη του Κοινοβουλίου που δίνουμε στην Κομισιόν τα μέσα, αλλά τα χρησιμοποιούν μόνο κατά των φερών, ε, αλλά όχι κατά της Ισλανδίας. Ε, ξέρω πολύ καλά τους Ισλανδούς και μας είπαν σαφώς ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν άποψη. Και αν ήμουν Ισλανδό, μπορεί και εγώ να έκανα τα ίδια. Αλλά πρέπει να δράσουν υπεύθυνα. Επειδή αυξήθηκαν τα συνολικά αλλιεύματα, πήγαμε 550 σε ένα εκατομμύριο. Αυτό σημαίνει ότι φέτος θα είμαστε στι 750.000 τόνου. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε με αυτή την τακτική. Φυσικά πηγαίνουν και οι κινέζικα σκάφη. Τι προσθέτουμε. δεν ε, ωφελείται τίποτα. Δεν ωφελείται η οικονομία μας. Απλώς παίρνουν τα ψάρια μας. Και δεν ξέρουμε πως υπάρχει αλλαγή σημαία. Δεν ξέρουμε από ποιες χώρες. Θα έπρεπε να ξέρουμε. Δεν αρκεί να λέμε δεν ξέρουμε τι σημαία φέρουν. Πρέπει να πούμε ότι τα μέτρα που θα εφαρμόσουμε δεν θα έχουν καμία επίπτωση. Όπως γράψαμε και στην έκθεσή μας, αυτό θα έχει επιπτώσεις και για το σαβρίδι και για αυτά που τρώνε οι σολομοί. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε πιο αποφασιστικά μέτρα. Εάν εφαρμόζαμε αυτά τα πιο αποφασιστικά μέτρα, θα επανέρχονταν στην Τράπεζα των Δεπραγματεύσεων. Ευχαριστώ την Επιτροπή που μας έκανε μια καλή επισκόπηση και φυσικά οι επικρίσει που δεν αφορούν το άτομο που μας παρουσίασε ε, την άποψη της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα νομίζω ότι συζητήθηκε αρκετά. Μία ή δύο ερωτήσει. Επειδή τροποποιήσαμε την ημερήσια διάταξη, είναι αλήθεια ότι να αρχίσουμε για τα Κανάρια στι 3 ε, που δεν θα το συζητήσουμε πολύ και η επόμενη έκθεση είναι στις 4.30 σημαίνει πως ε, δεν θα αξιοποιήσουμε καλά το χρόνο μας θα μπορούσαμε να περάσουμε κάποιο άλλο θέμα πριν τις 4.30. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να έρθουν κάποιοι μόνο με βάση την ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό προτείνω να αρχίσουμε στις 4, όχι στις 3, για να μην είμαστε μια ώρα περιμένοντας. Αν κάποιο θέλει να πάει μπροστά κάποιο θέμα του, να προταχθεί κάποιο άλλο θέμα, εντάξει. Αλλά επειδή δεν βλέπω κάτι τέτοιο, να αρχίσουμε με τα Κανάρια στις 4 και στις 4.30 θα έχουμε την παρουσίαση της έκθεσης, εντάξει. Θυμάστε ότι αλλάζουμε αίθουσα το απόγευμα δυστυχώ και πηγαίνουμε στην αίθουσα PHS 07 σε 50. Είναι αρκετά μακριά. Η κυρία Λοβίν. Για την ημερήσια διαταξία ξεπλάγιν που η παρουσίαση των επιδοτήσεων είναι μόνο μισή ώρα. Είναι επαρκής χρόνος συζήτησης. Ε, έτσι το προγραμμάτισε η γραμματεία. Όλα αυτά είναι πάντα κάπως σχετικά. Μετά υπάρχουν τρία θέματα που μπορεί να μας πάρουν περισσότερο χρόνο. Θα μπορούσαμε να προτάξουμε ένα για να ξεκινήσουμε στις τρεις. Αλλά όπως σας είπα, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα να γίνει. για το θέμα της Ταϊλάνδης θα έρθουν ε, άλλα άτομα απ' έξω. Άρα δεν έχει έννοια να έρθουν και να δουν ότι έχει ήδη συζητηθεί και το ίδιο νομίζω ισχύει για την έκθεση της κυρίας Λοβίν και για τα επιθετικά είδη. Μας είπαν ότι οι υπεύθυνοι από την Επιτροπή ε, ήθελα να έρθουν άλλη ώρα αλλά δεν είναι γενικά δυνατό θα προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε δεν υπάρχουν πολλές άλλες δυνατότητες ευχαριστώ πολύ σε άλλη αίθουσα